Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Περιμένοντας να έρθουν και τα άλλα μέλη του Κοινοβουλίου, λέω να αρχίσουμε γιατί έχουμε πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη και έχουμε ακροάσει για πολύ λεπτά και δύσκολα θέματα. Στα πρώτα πέντε λεπτά λοιπόν να σας ενημερώσω για τη συνεδρία των συντονιστών που είχαμε χθε όσον αφορά το μελλοντικό πρόγραμμα και ε, να σας πω τι αποφάσεις πήραμε. Όσον αφορά τις διαδικασίες για τον διορισμό των ε, ε, εισηγητών, απαλλαγή Λιμπεράσκη, 2010 ε, τώρα για τους ε, οργανισμούς, είναι υπεύθυνο το ΕΛΚ, Λοιπόν, ε, έχουμε επίση ε, το, τη διαδικασία Όμνιμου και το Ευρωπαϊκό και το Ελεκτικό Συνέδριο. Και όσον αφορά το Β, ε, θα ακούσουμε τα αποτελέσματα και θα έχουμε τον κύριο Λένε, πρόεδρο τη συνδιάσκεψη των πρόεδρων των Επιτροπών και έχουμε προθεσμία τη 29 Ιανουαρίου την Παρασκευή. Επιβεβαιώθηκε επίση η αντιπροσωπεία για την επίσκεψη στην Ελλάδα 27-29 Απριλίου. Η πρώτη από τι επισκέψει που θα κάνουμε θα είναι αυτή. Thank Μάλιστα, να μιλάω πιο αργά, ε, λέει ο πρόεδρος. 27 με 29 Απριλίου του 2010 και η γραμματεία αναλαμβάνει να διαλέξει το κατάλληλο ξενοδοχείο για το κατάλημα των μελών του Κοινοβουλίου. Εγκρίναμε επίσης την ακρόαση για τη διαφάνεια των διαθετικών ταμείων με τον κύριο Λιμπεράτσκι εισηγητή, ακολουθώντας την πρότασή του να ε, έχουμε και την ε, ε, ακρόαση για τη ΣΥΠΑ, δίνοντας όμως την Ευρωπαϊκή Διάσταση 13 Ιουλίου 2013 είναι η ημερομηνία. Τώρα, όσον αφορά την επίσκεψη στην Όλαφ για τις 4 Δευτέρου 2010 προς το παρόν αναβάλλεται περιμένοντας κυρίως να διατυπωθεί η γνωμοδότηση που ζητήθηκε από τις νομικές υπηρεσίες της Επιτροπής σε σχέση με ε, ε αυτό το κενό που υπάρχει στις υπηρεσίες της Όλαφ και με, την, ε, και με το διορισμό του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ε, τώρα, όσον αφορά τις ακροάσεις για το προσωπικό Όλαφ, θα γίνουν μετά από την παρουσίαση εκ μέρους του Επιτρόπου του σχεδίου και του προγράμματος εργασίας σε σχέση με την Όλαφ. Στη συνέχεια, ζητήσαμε από τις αστυνομικέ υπηρεσίες να απαντήσουν ως τον πιο γρήγορα στο θέμα αυτό του καινού, της κοινή θέση που υπάρχει στην Όλαφ για να δούμε ε, πώς ε, θα λάβουμε υπόψη τις απόψεις των πολιτικών ομάδων και να εξετάσουμε ε, την, ε, την νομιμότητα αυτή της θέσης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τώρα, όσον αφορά την απαλλαγή, να σας πω το εξή. Όσον αφορά το τμήμα το οποίο αφορά την Όλαφ, για το οποίο θα γίνει και εισαγωγική και η παρουσίαση στο Γενικό Γραμματεία, εδώ πρέπει να πω ότι ε, η συνεδρίαση ε, πάντα ε, γίνεται κλεισμένο των θυρών. Και υπενθυμίζω το παράρτημα 8 όσον αφορά ακριβώς τον, τον το απόρριτο χαρακτήρα αυτών που θα συζητηθούν στην ελόγω συνεδρίαση. Ε, θα, θα συμμετάσχουν, όπως αναφέρθηκε, μόνο τα μέλη του Κοινοβουλίου ή υπάλληλοι της Γραμματείας του Κοινοβουλίου, των οποίων η παρουσία είναι, θα κρίνεται ε, χρήσιμη ανάλογα με το θέμα της ημερής διάταξη και Πρέπει να σας πω επίσης ότι, ότι αποφασίστηκαν οι ακροάσεις των μελών του ελεκτικού συνεδρίου, των οποίων βεβαίω τα ονόματα θα επιβεβαιωθούν για τις ημερομηνίες 15 και 16 Τρίτου του 2010. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα το ποσό του προπολογισμού για την Επιτροπή όσον αφορά τις μελέτες του 2000, μελέτη του 2010. Ε, λίγο παραπάνω από 300.000 είναι το ποσό αυτό και μέσα στις ε, προσεχείς ημέρες θα εγκριθούν οι μελέτες που θα αποτελέσουν αντικείμενο χρηματοδότησης. Επίσης, να σας πω ότι αποφασίσαμε να αποστείλουμε επιστολή στον πρόεδρο της συνδιάσκεψης των Προέδρων, στον κύριο Λένε, για να αναφερθούμε στο γεγονός ότι η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα πρέπει πάντα να, ε, ε, να δίνει την άποψή της όσον αφορά το δημοσιονομικό κανονισμό Τη εξωτερική υπηρεσία που θα αρχίσει να λειτουργεί μετά τη Λισαβόνα. Το έχουμε πει επανειλημμένα και πιστεύουμε ότι ο ρόλο τη Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού θα πρέπει ε, να ε, είναι σημαντικός ακόμα από, την, από το στάδιο της μελέτης ε, της λειτουργίας αυτού του νέου οργάνου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένωσης. Επίσης αναφέρθηκε και ένα άλλο θέμα που αφορά την Επιτροπή και τη Γερμανία όσον αφορά ε, το, το ελεκτικό συνέδριο ε, και μέχρι την 28 Ιανουαρίου οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων θα πρέπει να ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους σε σχέση με μια παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα σε αυτή τη διαδικασία που ήδη έχει ξεκινήσει. Οι συντονιστές επίσης συμφώνησαν για τη διοργάνωση μιας συνεδρίασης Μόλις θα υπάρξει, ε, μόλις θα αναλάβει τα καθήκοντά της ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και, και, και, και προκειμένου ο νέος επίτροπος για να συζητήσουμε το θέμα αυτό που αφορά το νέο επικεφαλή Σόλαφ. Λοιπόν, αν δεν έχετε παρατηρήσεις, να πάω τώρα στο πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης που θα συζητήσουμε σήμερα και που αφορά την απαλλαγή 2008 Γενικός Προϋπολογισμός, τμήμα 3 Επιτροπή. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω όλους και να καλωσορίσω ιδιαίτερα την Επίτροπο Φερέρα Βάλτνερ. Να δώσω λοιπόν αμέσως το λόγο στον εκπρόσωπο του ε, Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, στον κύριο Μάρτιν Εκβίντα. Έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα κάνω μία σύντομη εισαγωγή στο 8ο κεφάλαιο της ε, ε, ετησίας εκθέσεως ε, του ελεγκτικού συνεδρίου. Όπως ξέρετε δημοσιεύουμε αυτή την έκθεση τον Νοέμβριο του 2009 και εδώ ασχολούμεθα με την εξωτερική βοήθεια, την ανάπτυξη και τη διεύρυνση. Επιπλέον το ε, συνέδριο έχει ε, διαμορφώσει έξι εκθέσεις μεταξύ από το, από το Ιανουαρίου 2009 καταρχήν σχετικά με τη διεύρυνση και τα θέματα νέας γειτονίας ιδίως για την Τουρκία, τα Δυτικά Βαλκάνια, τη Λευκορωσία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Δεύτερον, αναπτυξιακή βοήθεια σε ε, υγειονομικές υπηρεσίες στην υποσαχάριο Αφρική και το θέμα της αποτελεσματικότητας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της σχετικής βοήθειά της μέσω των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον στην έκθεση αυτή υπάρχει μία συνέχεια και παρακολούθηση ε, σχετικά με την, ε, έκθεση, την ειδική έκθεση 5 κάθετος 206 σχετικά με το πρόγραμμα ΜΕΝΤΑ για την Νότιο Μεσόγειο. 6,2 δισεκατομμύρια ε, δαπανήθηκαν συνολικά στο 2008 εκ των οι εξωτερικές σχέσεις και η ανάπτυξη ε, η αναπτυξιακή βοήθεια αναφέρονται στα 2 τρίτα περίπου των δαπανών αυτής της ε, πολιτικής. Τα υπόλοιπα καλύπτουν τη διεύρυνση 27% δηλαδή μεταβατικά μέσα και βοήθεια για την κατάρτιση θεσμικών οργάνων και ανθρωπιστική βοήθεια. Τα περισσότερα από τα έξοδα αυτά την χάνουν τις διαχειρίσεις από τρεις γενικές διευθύνσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Γενική Διεύθυνση για Ανθρωπιστική Βοήθεια ΕΚΟ, το Europe Aid για τις εξωτερικές σχέσεις και τα προγράμματα ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Διεύρυνσης για τις υποψήφιες χώρες. Επιπλέον τα έξοδα είναι, έχουν ε, διατεθεί επίσης και από τα Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Ταμεία. Ένα μεγάλο μέρος των δαπανών αυτών διαχειρίζεται, διαχειρίζονται αντιπροσωπείες Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις χώρες όπου χρηματοδοτούνται τα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οργανώσεις οι οποίες εφαρμόζουν τα προγράμματα μπορεί να είναι είτε διεθνείς οργανώσεις ή τοπικές και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις ή και κυβερνητικά κλιμάκια. Μέρος της αναπτύξεως και της βοηθείας δίδεται σαν ε, δημοσιονομική στήριξη υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Κύριε Πρόεδρε, το συνολικό συμπέτρασμα του ελεγκτικού συνεδρίου είναι ότι οι ε, συναλλαγές στον τομέα αυτό έχουν γίνει με σημαντικό επίπεδο λάθων ε, ε, και τακτικότητα εκ των οποίων ε, μόνο ένα μέρος ήταν ε, αποτελεσματικό, δηλαδή δεν υπήρχε μία τακτικότητα πληρωμών εξασφαλισμένη. Θα σας εξηγήσω λοιπόν ποια ήταν τα βασικά ε, σφάλματα τα οποία διαπιστώσαμε. Καταρχήν σφάλματα της επιλεξιμότητας, ιδίω όσον αφορά τις προϋποθέσεις για τα έξοδα και συμπερίληψη του ΦΠΑ και άλλο μη επιλεξίμων φόρων. Δηλαδή τα, τα παραστατικά τα οποία μας υποβλήθηκαν, τα τιμολόγια, οι αποδείξεις και ε, τα ε, ε, τραπεζικά οι τραπεζικοί λογαριασμοί δεν μας προσκομίστηκαν και δεν έγιναν σεβαστές οι χρονικές χρονικές προθεσμίες που είχαμε ε, ε, καθορίσει. Επίσης η διαδικασία για τους δημόσιους διαγωνισμούς παρουσίαζαν προβλήματα. Για τη Eurobaid το θέμα των ελέγχων στα κεντρικά αποτελεί, ε, είναι ένα αποτελεσματικό θέμα αλλά σε επίπεδο αντιπροσωπιών υπάρχουν αδυναμίες οι οποίες έχουν ιδίω σχέση με τους τους ελέγχους ε, σχετικά με ε, τις δημόσιες ε, επενδύσεις και τα συμβόλαια. Όσον αφορά τη Γενική Διεύθυνση ΡΕΛΕΞ διαπιστώσαμε πολλές αδυναμίες στους ελέγχους εκ και οι αδυναμίες σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση και την εποπτεία της ε, ε, οικονομικής πληροφόρησης όσον αφορά τα προβλήματα. Η Γενική Διεύθυνση ε, παρουσίασε αδυναμίες ή σε τη δυνατότητα εσωτερικού ελέγχου και στους ελέγχους εκ Post. Άλλωστε διαπιστώσαμε σημαντικές αδυναμίες ε, τόσο όσον αφορά τη διαχείριση των ε, ε, κεφαλαίων του προγράμματος ΦΑΡ στη Βουλγαρία. Καταλήγοντας, θεωρώ ότι για να βελτιωθεί η κατάσταση θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου εξάντε της Κομισιόν για τις πληρωμές και τα συμβόλαια Europaid και DG Relex Επίσης θα πρέπει να δοθεί περαιτέρω βοήθεια στις οργανώσεις που εφαρμόνουν τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως διεθνείς οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις και κυβερνητικά κλιμάκια και θα έπρεπε να υπόκεινται σε στενότερη παρακολούθηση. Και τρίτον, οι έλεγχοι και ε, ιδίω εκ των υστέρων θα πρέπει να προγραμματίζονται πιο ρεαλιστικά και να παρακολουθούν και τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών θα πρέπει να καταγράφονται και να αναλύονται συστηματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας ε, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ε, και τώρα πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Λιμπεράτσκι, να ζητήσω από την Επίτροπο Φέρερο να αν θέλει να το τοποθετηθεί σύντομα. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σιγητά, κυρίες και κύριοι μέλη της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι του Ελεκτικού Συνεδρίου. Ήρθα ενώπιόν σας σήμερα για να σας παρουσιάσω πράγματι τα αποτελέσματα των ε, προσπαθειών που συγκεντρώθηκαν στον τομέα των εξωτερικών δράσεων, έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη διαχείριση των κοινοτικών ταμείων και επίσης για να απαντήσω σε ερωτήσεις σας μετά από την ετήσια έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου που μόλις ακούσαμε. Κάτι τη διάρκεια της θητείας μου, διαρκώς προσπαθούσα να πετύχω ε, τα σημαντικά κονδύλια τα οποία μας έχετε εμπιστευτεί να αποτελούν αντικείμενο διαχείριση ώστε να τον καλύτερα, μερικέ φορέ κάτω από δύσκολε συνθήκε, σε πλήρη συνεργασία με του εταίρου μα. Στα πλαίσια αυτά, η βελτίωση τη συνεργασία μα με τα Ηνωμένα Έθνη αποτελεί ένα θέμα το οποίο μα απασχόλησε σε μεγάλο βαθμό λάβαμε υπόψη στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη παρατηρήσεις σα και το 2009 συνάψαμε συμφωνία για τα για ε, τους, ε, τους πρότυπους όρους αναφοράς για τις αποστολές επαλήθευση που προστίθενται στα μέτρα τα οποία ήδη ελήφθησαν τα προηγούμενα χρόνια με τα Ηνωμένα Έθνη όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές σε θέματα ορατότητας καθώς επίσης ε, και στην δημοσιονομική παρακολούθηση των κονδυλίων μας. Η ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου σχετικά με την σύνδρομή μας, όπως εφαρμόστηκε από τον ΟΗΕ και που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, υπογραμμίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Ταυτόχρονα όμως αναφέρεται σαφώς ότι πρέπει να σημειωθεί ακόμα μεγαλύτερη πρόοδος, κυρίως όσον αφορά ε, τις εξηγήσεις που θα πρέπει να δοθούν για την επιλογή να καταφύγουμε στους ε, οργανισμούς των ΗΕ ή όσον αφορά την πρόσβαση και το περιεχόμενο των εκθέσεων των ΗΕ κατά τις, ε, τα στάδια ελέγχου. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να μελετήσουμε πολύ μεγάλη προσοχή τα συμπεράσματα του συνεδρίου και να λάβουμε τα απαραίτητα ε, συμπληρωματικά μέτρα με βάση των ε, υποδείξεων. Τώρα κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στο, ε, στην ουσία της συνδρομής μας που αποτελεί που αντιπροσωπεύει το 80% της συνολικής μας εξωτερικής βοήθειας και για το μεγαλύτερο μέρος υλοποιείται απευθείας από τις αντιπροσωπείες μας. Καταρχήν σημειώνουμε ότι στη γενική του έκθεση το συνέδριο σημείωσε ότι υπήρξαν βελτιώσει όσον αφορά τα συστήματα ελέγχου και εποπτείας, ακόμα και αν και φυσικά αυτό ε, είναι, και είναι φυσικό βεβαίως να ε, πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειές μας σε ορισμένους τομείς. Βεβαίω αντιλαμβανόμαστε καλά τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν ορισμένοι οι οποίοι προσπαθούν να λάβουν υπόψη τους κανόνες μας και τις απαιτήσει μας που πάντα είναι λεπτομερείς και μερικές φορές είναι πολύπλοκοι έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ο καλός κίνδυνος και να ο καλός, ε, η καλή διαχείριση συγγνώμη, και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος. Για να τους βοηθήσουμε και εμείς, το EuroPay τώρα εργάζεται με βάση ένα χρηματοπιστωτικό, ε, ένα, ένα, ένα kit, ε, ένα toolkit, ένα kit εργαλείων για τη χρηματοπιστωτική διαχείριση, το οποίο έχει στόχο να βοηθήσει οργανώσεις όπως οι μη οργανώσει οργανώσει να διαχειρίζονται τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι μέρο από τη λύση του προβλήματο θα βρεθεί στην περαιτέρω απλοποίηση των κανόνων και των διαδικασιών. Παράλληλα, αναλάβαμε σημαντική δέσμευση τα τελευταία χρόνια για να προωθήσουμε την οικοδόμηση εσωτερικών ε, δυνατοτήτων ε, στι χώρε εταίρου και εμπνευστήκαμε σε μεγάλο βαθμό από την εργασία ε, του συνεδρίου στην ειδική έκθεση για την τεχνική αρρωγή. Ταυτόχρονα σημειώσαμε πρόοδο σε ένα σημαντικό τομέα που τον τονίζει το συνεδρίο τα πρόσφατα χρόνια, δηλαδή στην κάλυψη του ελέγχου ε, και τη χρήση των συμπερασμάτων των ελέγχων. Βελτιώσαμε τη μεθοδολογία του ελέγχου με νέου πρότυπου όρου αναφορά για του διάφορου ε, τύπου ελέγχου και για μια διαρκή και συνεπή ανάλυση κινδύνου. Πιστεύω ότι υπήρξε σημαντική πρόοδο όσον αφορά και την ποσότητα αλλά και την ποιότητα του εξωτερικού ελέγχου τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, το 2008 υπήρξε αύξηση κατά 37% όσον αφορά τον αριθμό των ελέγχων της Europaid που ολοκληρώθηκαν και αυτό σε σύγκριση με το 2007. Το ίδιο ισχύει και για τους ελέγχους του Ρέλεξ. Όλα τα ωφέλη από αυτή την εργασία μπορεί να μην είναι ακόμα ορατά, διότι απαιτείται κάποιο χρόνο για να αποδώσουν καρπί τα συγκεκριμένα μέτρα. Και βεβαίω αντιλαμβάνομαι και κατανοώ ότι ο ρόλο του συνεδρίου είναι να μα ενθαρρύνει έτσι ώστε να έχουμε ακόμα καλύτερε επιδόσει το, η ανάλυση κόστου ωφέλου των ελέγχων, που επίση τόνισε το συνέδριο, αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο η Επιτροπή το λαμβάνει υπόψη ιδιαίτερα σοβαρά. Πέρυσι, ο Συνάδελφο μου Σιμ Κάλλα και οι υπηρεσίε του ήδη ξεκίνησαν την εργασία για μια ε, ανάλυση σε βάθο κόστου ωφέλου όσον αφορά τρει από, τις, τομεί πολιτική πολιτική τομείς ε, πολιτικής την εξωτερική δράση. Η Επιτροπή θα συμποβάλει έκθεση του χρόνου με βάση τα ευρήματα αυτά. Τέλος, επειδή κύριε Πρόεδρε, είναι η τελευταία φορά που μου δίνετε ευκαιρία να, έρχο, να εμφανίζομαι ενώπιον σα με την ιδιότητά μου τη Επιτρόπου, θα ήθελα για άλλη μια φορά να σα ευχαριστήσω όλου για τη συνεργασία σα και επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και το ελεκτικό συνέδριο για την επικοδομητική του προσέγγιση. Θα ήθελα να είστε βέβαιοι ότι κατέβαλα κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη διαχείριση των εξωτερικών κονδυλίων βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένω τώρα τι ερωτήσει σα. Εγώ σας ευχαριστώ, Επίτροπε. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Λιμπεράδης και τον εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να τονίσω καταρχήν ότι υπάρχει μεγάλη βελτίωση όλα αυτά τα χρόνια διαδοχικά της απαλλαγής. Παρόλα αυτά το ποσοστό σφαλμάτων είναι εντυπωσιακό. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν. Κυρία Επίτροπε, Καταρχήν να δούμε τις ερωτήσεις ε, που αφορούν τις ε, μακρές καλές συστάσεις που ακόμη δεν έχουν ε, ληφθεί υπόψη, όπως δείχνουν τα έγγραφα. Πρώτα απ' όλα, ένα follow-up των συστάσεων, ορισμός επιδόσεων, που θα επιτρέπει αποτελεσματικό αντίκτυπο των επιπτώσεων. Ακόμη δεν έχουν ε, υπάρξει στρατηγικοί στόχοι και δίκτες ε, απόδοσης σε όλα τα έγγραφα. Οπότε, ερωτώ, τι κάνει η Κομισιόν για να ανταποκριθεί στη σύσταση του συνεδρίου ε, για τις συστάσεις, της ορθές και της μακράς διάρκειας. Αυτά καταρχήν και μετά θα ακολουθήσουν και άλλες ερωτήσεις. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Εισηγητά, πράγματι το έγγραφο εθνικής στρατηγικής αποφασίζεται για, μια, για κάθε χώρα και προβλέπει συνολική περιγραφή της κατάστασης στη χώρα. Παρουσίαση τους τομείς ε, στρατηγικής προτεραιότητας για παρεμβάσεις, ώστε να αντιμετωπίζονται οι μεγαλύτερες προκλήσεις που εντοπίζονται στη χώρα, όπως και μια παρουσίαση των βασικών στόχων και δικτών αποτελεσμάτων και αντικτύπου. Τώρα, σύμφωνα με τον κανονισμό ENPI, η αρχική κατάσταση και η τελική αξιολόγηση με βάση τους δείκτες που αναφέρεται προσδιορίζονται αργότερα σε μετέπειτα στάδιο όταν καθορίζονται τα προγράμματα δράσης τη στιγμή της διατύπωσης του προγράμματος όταν ε, τότε ορίζονται οι στόχοι του προγράμματος ε, λεπτομερώς και υπάρχουν και δείκτες πλέον οριστικοί σε συνεργασία με ε, δωρητές ε, ή άλλες χώρες και χρησιμοποιούνται για να παρακολουθήσουμε τη φάση της υλοποίησης και χρησιμοποιούνται και στην αξιολόγηση εξ η Κομισιόν εξέτασε το θέμα ούτως ώστε να προσδιορίσει δείκτες καλύτερους, κατάλληλους, κατά τη διατύπωση των προγραμμάτων, των ειδικών προγραμμάτων, των projects. Και υπάρχει και ένας ε, καινούριος οδηγός για τη χρήση τους, ούτως ώστε να γίνονται οι μετρήσεις της ε, απόδοσης. Αυτό ολοκληρώνεται τώρα και θα οριστικοποιηθεί αυτός ο οδηγός ε, το 2010, το πρώτο εξάμεινο. Αυτός ο οδηγός υπογραμμίζει τις αναλύσεις και τις ικανότητες των χωρών σε συνεργασία με άλλες χώρες εταίρους εις ό,τι αφορά τους δείκτες ανταπόκρισης και απόδοσης. Σας παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Τώρα, για την ε, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εξωτερικής πολιτικής της Κομισιόν. Η Κομισιόν πώς ε, εντοπίζει υψηλού κινδύνου περιοχές, πώς τις ε, προσεγγίζει, τα συστήματα ελέγχου για αυτά τα κονδύλια πώς χρησιμοποιούνται, γιατί πρέπει να προσδιοριστούν διαφορετικά επίπεδα κινδύνου στις διάφορες περιοχές του κόσμου ε, και είναι μια ευρία γκάμα αυτή. Τι αποτελεσματικότητα έχουν τα συστήματα ελέγχου και κατά τη γνώμη σας έτσι αυξάνεται η θετική στάση και το θετικό κλίμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τα κονδύλια που παρέχουμε. Ευχαριστώ κύριε Ισηγητά. Είμαι ευγνώμων μάλιστα για την ερώτηση γιατί νομίζω ότι ε, αφορά το πραγματικό πολιτικό αντίκτυπο της ε, ε βοήθειας σε περιοχές κρίσης. Πολλές φορές ε, δεν είναι αυτές συνήθεις χώρες όταν υπάρχει κρίση δεν πάνε όλα ομαλά, το περιβάλλον είναι υψηλού ρίσκου και ακριβώς αυτή είναι και η πρόκληση της εξωτερικής βοήθειας. Οι περισσότερες χώρες εταίροι μας πρώτα απ' όλα έχουν ε, αναποτελεσματικά, δημοσιονομικά και διοικητικά συστήματα που πρέπει να μεταρρυθμιστούν και να ενισχυθούν, να βελτιωθούν με προγράμματα εξυγχρονισμού και δημιουργίας ικανοτήτων. Κατά δεύτερο λόγο υπάρχει ως επιτοπλίστων πολιτική αστάθεια και πολύ συχνά και συγκρούσεις που ξεπερνούν το σύνηθες εργασιακό περιβάλλον μας. Επίσης υπάρχει συχνά ε, μεγάλη φτώχεια και διαφθορά. Αυτά ε, συνδυάζονται ως παράγοντες στις πιο φτωχές χώρες όλα μαζί ως εκ τούτου πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν διαχειριζόμεθα εξωτερική βοήθεια. Γι' αυτό η Κομισιόν ε, και κατά το παρελθόν και στο μέλλον κάνει πολλά, ε, εφαρμόζει πολλά μέτρα ελέγχου για να αντιμετωπίσει τους διαφορεοποιημένους και πολλούς κινδύνους. Σε αυτό το τομέα σφάλματα κύριε Ισηγητά οπωσδήποτε που έχουν και δημοσιονομικές επιπτώσεις ενδεχομένως θα συμβούν. Δεν είναι τελείως ε, δυνατόν να τα αποφύγουμε. Τώρα τι συστήματα ε, ελέγχου υπάρχουν στο κεφάλαιο 8 της ετήσιας έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου, εκεί όπου το συνέδριο παρουσιάζει μια σχετικά ουδέτερη αξιολόγηση παρουσιάζει ένα επίπεδο σφαλμάτων 2 με 5% κατά μέσον όρο ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό σε αυτά τα πλαίσια να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Έτσι επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα της βοήθειας που πρέπει να αναβαθμιστεί με όλες τις μορφές. Τι κάνουμε λοιπόν. Αφενός θα ε, ε, γίνονται πάρα, πολλές, πάρα πολλοί έλεγχοι, επαληθεύσεις από εξωτερικούς ελεγκτές πέρα από αυτούς που γίνονται από τους δικαιούχους και τον εσωτερικό έλεγχο, γιατί έχουμε και υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Και επί τη βάση αυτών των εκθέσεων μετά αναλύονται τα αποτελέσματα, παρακολουθούνται τα πορίσματα, αποτελέσματα και αντλούνται και διδάγματα. Και μετά οι ελεγκτές αποστέλλονται για να κάνουν λεπτομερή προηγούμενη αξιολόγηση των συστημάτων ελέγχων των χωρών εταίρων και των διεθνών οργανισμών πριν αρχίσει η υλοποίηση της εξωτερικής βοήθειας, πριν δοθούν τα χρήματα. Και οι αντιπροσωπείες θα πρέπει να υποβάλουν ε, έκθεση πρόοδου κάθε έξι μήνες και να αναφέρονται συγκεκριμένα σε θέματα διαχείρισης. Η αποτελεσματικότητα λοιπόν των προτύπων εσωτερικού ελέγχου αξιολογείται ετησίως επίσης. Επίσης ε, έχουμε ε, επιτόπιες αποστολές επαλήθευσης που οργανώνονται κεντρικά για να εξετάσουν ε, πώς εργάζονται επιτόπου Και επίσης γίνονται και έλεγχοι των όλων των συναλλαγών που δείχνουν αυτές οι τελευταίες μετά την τελική πληρωμή χαμηλό ποσοστό σφαλμάτων. Γιατί καμιά φορά εξετάζονται οι προσωρινές ε, πληρωμές ε, στην αρχή και στο μέσον, στο τέλος είναι χαμηλό το επίπεδο ασφαλμάτων. Επίσης, ε, η παρακολούθηση του έργου του ελεγκτικού συνεδρίου λαμβάνεται υπόψη. Αυτός λοιπόν ο ενδεικτικό κατάλογος πηγών που ε, τροφοδοτούν τις υπηρεσίες μας δεν είναι εξαντλητικός, αλλά δείχνει πόσο προσεκτικά οι υπηρεσίες της Κομισιόν ενημερώνουν με σοβαρότητα για τις ετήσιες ε, δραστηριότητές τους και μας ενδιαφέρει να εργαζόμεθα ε, σε ένα σωστό επίπεδο και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη όλα τα, όλους τους κινδύνους που αφορούν τη λειτουργία και την διαχείριση των ε, κονδυλίων. Ωραία αυτά που μας λέτε, αλλά ο κύριος ανέφερε μεγάλα σφάλματα, κατηγορίες σφαλμάτων πολλές, όπως δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την πληρωμή, τη δαπάνη ή τη συμπερίληψη του ΦΠΑ αλλά και άλλα περιστατικά αναφέρονται με αποδείξεις, τιμολόγια, εξτρέ τραπεζών κλπ. κλπ. Αντιλαμβάνομαι ότι ο βασικός σας στόχος ήταν να εξυπηρετήσετε την ε, εξωτερική βοήθεια και να λάβετε υπόψη στο ελεγκτικό συνέδριο. Πώς μπορείτε όμως να εξηγήσετε αυτές τις κατηγορίες σφαλμάτων. Υπάρχουν αμέλειες, αδυναμίες, αδράνεια ή μήπως είναι δικαιολογημένα σφάλματα, δηλαδή ανεκτά, θεμητά να τα πούμε. Ε, αμέλειες, αδυναμίες, αδράνεια, ε, θεμητά σφάλματα. Θα ήθελα τη γνώμη σας πάνω σε αυτά τα σφάλματα, διότι είστε έμπειροι και υπεύθυνοι επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ κύριε εισηγητά. Πράγματι, όπως προείπα, σύμφωνα με το συνέδριο και εσείς αναφερθήκατε σε αυτό, ο δημοσιονομικός αντίκτυπος των σφαλμάτων το 2008 μετά τον έλεγχο του έτους αυτού είναι από 2 μέχρι 5% του δείγματος ελέγχου για δραστηριότητες που χρηματοδοτήθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό αλλά και τα Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά ε, τα κονδύλια του, του, Αμείου Ανάπτυξης. Το συνέδριο δεν εντοπίζει ε, τυπικά σφάλματα όπως ελείποντα ε, έγγραφα, ή ε, σφάλματα στις προκαταβολές ή στις ενδιάμεσες πληρωμές που μπορεί να πληρωθούν. Πολλές φορές ε, ε, μέχρι την τελική πληρωμή διορθώνονται αυτά. Εκεί διορθώνονται ήδη κάποια σφάλματα. Μετά την τελική πληρωμή δεν μπορεί να αποκατασταθούν τα σφάλματα. Έτσι λοιπόν αυτά τα σφάλματα έχουν, έχουν να κάνουν υποθέσεις που μπορούν τα ποσά να ανακτηθούν. Και στο EuroPaid του 2008 και τις ανακτήσεις ποσών 116 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με, ε, ε, με βάση τον κοινοτικό προϋπολογισμό εδώ συγκαταλέγονται όλα τα εντάλματα ανάκτησης όχι μόνο αυτά που προκύπτουν από σφάλματα ή μη δαπανηθίζεσες ε, δαπάνες κλπ. Αυτό αποτελεί καλή ένδειξη για το ποσό των μη επιλέξιμων ε, πληρωμών που περιλαμβάνονται στο ποσό αυτό. Έτσι λοιπόν συνολικά μπορώ να πω ότι καμιά φορά υπάρχουν διαδικαστικά σφάλματα πολύ περισσότερο από ό,τι σφάλματα που έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο. Λιγότερο από τα μισά από όλα τα σφάλματα που εντόπισε το συνέδριο σε εξωτερικές σχέσεις ε, προσδιορίζονται προσδιορίζονται ε, ποσοτικά οικονομικά. Τα περισσότερα σφάλματα δεν επηρεάζουν τον προϋπολογισμό της κοινότητας και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Βεβαίως ε, τα λάθη είναι ανθρώπινα, ουδής αλάνθαστος, καμιά φορά είναι αμέλεια, καμιά φορά εντοπίζουμε δυναμίες. άλλες φορές θα έλεγα ότι πρόκειται ακριβώς γι' αυτό ότι ε, οφείλονται στη διαδικασία κάποια σφάλματα που δεν έχουν όμως ε, δημοσιονομικό αντίκτυπο. Όμως ε, το συνέδριο έχει μια συνολική εικόνα. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε δύο τελευταίες ερωτήσεις πολύ σύντομες. Η πρώτη ερώτηση. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι οι σχέσεις εργασίας με τα Ηνωμένα Έθνη βελτιώθηκαν. Αυτό αποτελεί ένα επίτευγμα. Το γνωρίζω τι σημαίνει αυτό. Γιατί πραγματικά με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το δίκτυο ε, των Ηνωμένων Εθνών στι ε, ενδιαφερόμενε χώρε. Εξακολουθούν όμω να περιμένουν προβλήματα που δεν έχουν ακόμα επιληθεί. Θα ήθελα να ρωτήσω, εσεί Επίτροπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι πιστεύετε, ποιο είναι ο πιθανό τρόπο ε, με τον οποίο θα μπορούσαμε ε, να καταφέρουμε μια πραγματικά ομαλή συνεργασία. Εδώ πρόκειται για πολλά χρήματα για δύο ιδιαίτερα ε, σημαντικούς ε, διεθνείς οργανισμούς, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένα Έθνη και, και είναι σαφές ότι θα έπρεπε τα ενδιαφέροντά μας και τα συμφέροντά μας να είναι προς την ίδια κατεύθυνση, να είναι ευθυγραμμισμένα. Ευχαριστώ κύριε Σίγητα. Πράγματι, πρόκειται για μια ερώτηση, για ένα ερώτημα που μας έχει απασχολήσει εδώ και πολύ καιρό, πρέπει να το πω. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ε, από πολιτική άποψη η συνεργασία μας με τα Ηνωμένα Έθνη μέσω ε, των ε, ταμείων των, όλων των δωρητών μας επέτρεψε και θα επιτρέψει και στο μέλλον σε ορισμένες περιπτώσεις στην Επιτροπή να παρέμβουμε σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ορισμένες υποθέσεις όπου διαφορετικά θα ήμασταν, θα ήμασταν αποκλεισμένοι. Δηλαδή εκεί όπου έχει σταματήσει η συνεργασία ε, ή όπου διαφορετικά δεν ε, τίθεται θέμα νομιμότητας ε, ή όπου χρειαζόμαστε την ουδετερότητα της Παγκόσμιας Τράπεζας και των Ηνωμένων Εθνών. Να πω λοιπόν ότι μπορεί να μην είναι πάντα εύκολο να συνεργαζόμαστε με τους διεθνείς αυτούς οργανισμούς, και βεβαίως ε, παρόλα αυτά προσπαθούμε και έχουμε κάνει ε, μεγάλη πρόοδο. ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Παρόλα αυτά πάντως είναι κρίσιμη ε, εταίροι τα, οι διεθνείς οργανισμοί αυτοί για την ανάκαμψη στην περίοδο μετά από, τις, μετά από πολέμους συγκρούσεις. Προσπαθούμε ε, και οικονομικά και με, τους, με τις δομές προσπαθούμε ε, να πετύχουμε μια κατάσταση με βάση την οποία θα, μπορεί πάντα να λένε, θα μπορούν πάντα τα Ηνωμένα Έθνη να ε, αναφέρουν τη γνώμη τους και ε, να είμαστε και εμεί ε, και είμαστε, να είμαστε και εμείς σύμφωνοι με τι διεθνεί μας δεσμεύσεις σε επίπεδο αποτελεσματικότητα βοήθεια. βοήθειας. Γνωρίζω ότι το Κοινοβούλιο δεν ήταν πάντα ικανοποιημένο ή τουλάχιστον δεν ήταν απόλυτα ικανοποιημένο για τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε με αυτού του οργανισμού. Γι' αυτό πρέπει να σα πω ότι καταβάλαμε κάθε προσπάθεια για να δίδουμε, δίνουμε πληροφορίε στο Κοινοβούλιο για να ε, αντιμετωπίσετε κι εσεί τι ανησυχίε σα για θέματα όπω ορατότητα, διαφάνεια, συστήματα ελέγχου όταν δηλαδή ε, πρόκειται για διαχέτευση κονδυλίων μέσω συνεργασίας με εταίρους όπως οι διεθνείς οργανισμοί πληροφορίες για τους δικαιούχους των κονδυλίων που δημοσιεύονται από τις διεθνείς οργανώσεις από τους διαχειριστές των ταμείων της Παγκόσμιας Τράπεζας και των Ηνωμένων Εθνών. Ξέρω ότι τους έχουμε ζητήσει να έρχονται στο Κοινοβούλιο και να εξηγούν απευθείας εσά πώς, τι γίνεται με τα χρήματα αυτά και ε, ε, και βεβαίως να υπάρξει λεπτομερής επαφή με το, με το Ταμείο Όλων των Δωρητών όσον αφορά επίσης ε, την επαλήθευση των Ηνωμένων Εθνών των όρων αναφοράς, θέματα τα οποία έχουν αναφερθεί δημόσια και το πώς ερχόμαστε σε επαφή με τις αποστολές επαλήθευσης. Άρα, κύριε Σιγητά, και εμεί είμαστε έτοιμοι να δούμε το θέμα αυτό και να κάνουμε και προτάσει στα πλαίσια τη αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, γιατί σε παρελθόν δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να διαχειρίζεται αυτά τα, ε, τα, τα ταμεία ε, των πολλαπλών δωρητών, πράγμα το οποίο δεν μπορούσε να γίνει στο παρελθόν. Ε, αυτή τη στιγμή αυτά έχω να σας πω. Ευχαριστώ. Uh, και η τελευταία ερώτηση όσον αφορά την Βουλγαρία. Γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν παρατυπίες και ξέρετε ότι ε, έγινε, έγινε και αναστολή των, των πληρωμών. Επίτροπε, τι γίνεται με τη Βουλγαρία σήμερα, μπορείτε να μας πείτε. Ποια, γιατί ξέρουμε τη θέση του ελεκτικού συνεδρίου. Σα ζητώ συγγνώμη κύριε Σιγητά. Δεν είναι, δεν, δεν είναι τομέα εξωτερική δράση. Ε, η Βουλγαρία δεν, Μάλιστα, δεν θέλετε να απαντήσετε λοιπόν, κατάλαβα. Ωραία. Να πάρω λοιπόν, να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που έχω άλλη μια ερώτηση, να σας ρωτήσω. Τι, ποια θα ήταν η συμβουλή που θα μπορούσατε να δώσετε στον ε, διάδοχό σας, έτσι ώστε το επίπεδο σφάλματος να φτάσει σε ανεκτά επίπεδα. Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια έχετε έτσι μια συμβουλή να δώσετε στο, στον επόμενο επίτροπο. Εκτός μικροφώνου επίτροπος. Αυτό που ο Γενικός Διευθυντής μου, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, όλοι έχουν ξεκινήσει να ε, υπάρξει συνέχεια με, σε μια σοβαρή βάση. Γιατί έχουμε αντλήσει πολλά διδάγματα από την εμπειρία μας και θέλουμε να συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό ε, είναι το ένα. Δεύτερον, σε περισσότερο πολιτικό επίπεδο να σας πω το εξής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητήσουμε αυτό το ανεκτό, το μικρό επίπεδο σφαλμάτων στην εξωτερική δράση μα. Γιατί κοιτάξτε, για παράδειγμα, τι έγινε με την ΑΕΤ. Η ΑΕΤ είναι μια καινούργια υπόθεση. Όλοι είδαμε τι καταστροφέ ε, και ε, τα δεινά που υπέστη ο λαό τη ΑΕΤ. Μπορείτε να φανταστείτε όταν στο, στο μέλλον θα δώσει πολλά χρήματα και η Επιτροπή και τα κρατημέλη. Όλοι θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν το λαό της ΑΕΤ. Και αυτό απαιτείται. Αλλά πραγματικά πιστεύετε ότι εκεί με την διοικητική ικανότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή τα πάντα ε, θα ε, ε, διεξαχθούν ομαλά, μα δεν είναι δυνατόν. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό και αυτή αν θέλετε θα είναι η συμβουλή μου στον επόμενο επίτροπο, αλλά και στην επιτροπή σας, είναι να γίνεται μια αξιολόγηση με βάση τα συγκεκριμένα γεγονότα και να λέμε πρέπει να υπάρξει ένας ανεκτός κίνδυνος, μικρός αλλά Κοιτάξτε, εδώ δεν μιλάμε για τη Δανία ή για κάποιο άλλο κράτος μέλος. Ε, μιλάμε για άλλε χώρε, όπω η ΑΕΤ. Ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρο. Τώρα έχουμε άλλα 30 λεπτά. Έχουμε μια σειρά ομιλητών. Σα παρακαλώ και στι ερωτήσει και στι απαντήσει να είστε όλοι σύντομοι. Ο κύριο Χατζημακάρξ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Επίτροπο όχι μόνο για τις απαντήσεις σήμερα αλλά για όλες τις επιδόσεις της τελευταίας πενταετίας. Και τώρα μία άλλη κυρία θα συνεχίσει αυτή την εργασία. Εσείς θα ήσασταν πάρα πολύ καλοί σε αυτό και βοηθήσατε την Ευρώπη πάρα πολύ. Σας σεβόμαστε πάρα πολύ και ίσως ε, γι' αυτό ε, ε, εξεφράστη έτσι και το ελεγκτικό συνέδριο είναι κάτι το οποίο σημειώνεται διότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε είμαστε πάρα πολύ ευγενικοί μιλάμε για χρήματα των φορολογουμένων 6,2 ε, δισεκατομμύρια στο σύνολο και ε, τουλάχιστον αυτή τη φορά λέμε δεν κάηκε το κάηκε με το σπίτι μας έπιασε φωτιά αλλά σώθηκε το γαράζ κάτι τέτοιο βλέπουμε δηλαδή κάθε ε, μικρή επιχείρηση που αναλαμβάνεται. Παραδείγματο χάρη βοήθεια για τα παιδιά στη Γερμανία. Πρέπει να δώσουν, να απολογηθούν και να στείλουν τα αποτελέσματά τους. Γίνεται το ίδιο και για, τη Χαϊτή, για την Αϊτή. Και είτε μας γυρίζουν τα υπολοιπόμενα χρήματα με έμβασμα ή κάτι. Ξέρουμε ότι όλα δεν μπορούν να ελεγχθούν μέχρι την τελευταία τελεία. αντιλαμβάνουμε λοιπόν ότι ε, υπάρχει ε, μια αντιπαράθεση μεταξύ justified και tolerable, δηλαδή αιτιολογημένο ή ανεκτό. Διότι εμείς ε, κανονικά θα έπρεπε να ακολουθήσουμε αυτό που είπατε, να θέσουμε ένα όριο. Και θα ήθελα να ζητήσω από το ελεγκτικό συνέδριο να σκεφτεί την πρόταση αυτή. Αλλά αυτά τα οποία λέμε εδώ δυστυχώς είναι ουσιαστικά ουσιαστικά ξέρω ότι ο υπεύθυνο είναι πολύ ευσυνείδητος και Ολλανδός επιπλέον. Άρα είναι ένας καλός συνδυασμός. Αυτό που μας λέει λοιπόν είναι πολύ αξιοπρόσεκτο διότι είναι μια συζήτηση που κάνουμε μαζί του με το, μεταξύ Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Αναπτυξιακό Ταμείο όπου και εκεί υπάρχουν αδιάφανοι τομείς. Και στο τέλος οι Ευρωπαίοι και εσείς με διαφορετικό καπέλο στο μέλλον βλέπετε ότι μιλάμε για διασπάθηση των ευρωπαϊκών δημοσίων πόρων. Ε, αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε, γι' αυτό και για το μέλλον θα ήθελα να σας παρακαλέσω να πείτε στην ε, κυρία που θα σας διαδεχτεί ε, τι συζητήσαμε διότι βεβαίως η Γενική Διεύθυνση θα παραμείνει. Οι κύριοι που εκπροσωπούνται εδώ σήμερα θα παραμείνουν και κάποια στιγμή και εμείς θα καταφέρουμε καλύτερα. Ε, ε, ε, βλέπουμε ότι ο κύριος Μπαρόζο χρησιμοποιεί την αρχή διέρη και βασίλευε όλο και περισσότερο. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να έχουμε μία ενιαία αντιμετώπιση και να υπάρχει ένας μοναδικός επίτροπος υπόλογος. Και εδώ ε, εδώ ανοίγω μια παρέανθηση ευτυχώ που δεν το ανέλαβε η κυρία Γέλεβα την οποία δεν θεωρώ ότι θα ήταν ε, αρμόδια κλείνω την παρέθεση είμαι αντικειμενικό, αλλά ήταν ακατάλληλη αυτό το οποίο θα αλλάξει με την Lady Ashton διότι εσείς δώσατε ε, μία συμβουλή για το τι θα έπρεπε να προσέξει τι θα αλλάξει όμω, γιατί αυτή θα παίξει ένα συντονιστικό ρόλο μπορούμε να αναμείνουμε ότι όταν θα την ακούσουμε ε, σαν ε, ε, επόμενη υπεύθυνη θα ακούσουμε ότι υπό το συντονισμό της θα υπάρχει καλύτερη δρομολόγηση των θεμάτων για να το πω στη γλώσσα σας. Καταρχήν, σας ευχαριστώ κύριε ε, Ευρωβουλευτά για τον τρόπο που απευθυνθήκατε απέναντί μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Όντως τα πέντε χρόνια αυτά ήταν πολύ έντονα και ευχαριστώ για την αξιολόγησή σας. Κατά δεύτερον λόγον, ακόμη και αν το ελεκτικό συνέδριο μιλάει για 2-5% αντικειμενικό λάθος πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του τι συμβαίνει συχνά στο διαδικαστικό και τελικά των θεμάτων που έχουν οικονομικές επιπτώσεις. Δηλαδή και αυτό θα μπορέσουμε να αμφισβητήσουμε και ουσιαστικά να εστιαστούμε σε αυτό το οποίο έχει χρηματικές επιστώσεις διότι τα υπόλοιπα έχουν σωθεί εντωμεταξύ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί έχουν γίνει έλεγχοι. Καθ' όλη τη διαδικασία λοιπόν και το ε, υπεστήριξα, ευχαριστώ για τη βοήθειά σας, ε, είναι βασικό να γίνει μία ανάλυση με το χέρι στην καρδιά, κατά τρόπον ώστε να μπορούμε να πούμε αυτό το πράγμα δεν έχει νόημα. Υπάρχουν τόσοι έλεγχοι που εγώ πολλές φορές αναρωτιέμαι, όπως το είπαν και άλλοι, πώς είναι δυνατόν το επιτελείο μου να μπορεί να εργάζεται εξάντε, εξ post, procurement, όλοι οι έλεγχοι, ε, εξωτερικοί, οι Όλαφ, όλοι και όλα αυτά πρέπει να γίνουν στο ποδάρι πάρα πολύ γρήγορα. Πολλές φορές τετραγωνίζουμε τον κύκλο και θα ήθελα παρακαλώ αυτό να το λάβετε υπόψη σας. Είμαι η τελευταία η οποία δεν ήθελε, ε, η οποία, είμαι πάντοτε αυτή η οποία ήθελε να δουλεύει σωστά και νομίζω ότι το πέτυχα και για μένα και για το προσωπικό μου. Ε, πρέπει να σας πω ότι όσο με αφορά σκέφτηκα ποια θα μπορούσε να είναι η κατανομή. Βεβαίως εγώ μπορούσα να πω στον πρόεδρο μόνο την προσωπική μου γνώμη, αλλά η γνώμη μου ήταν σαφής. Δηλαδή ότι έπρεπε ε, να υπάρχει ε, μία ε, επίτροπος γυτνιάσεως, διότι η πολιτική γυτνιάσεως είναι πολύ σημαντική και η Lady Άστον δεν μπορεί να τα καλύψει όλα. Ξέρω ότι εγώ κάλυψα ένα μέρος των λειτουργιών ε, αλλά υπήρχε και ο Σολάνα ο οποίος έκανε τα υπόλοιπα δεν μπορεί ένας άνθρωπος να τα κάνει όλα δεν είναι υπεράνθρωπος πρέπει οι άνθρωποι να μπορούν να μπουν και στις λεπτομέρειες και κάποιος πρέπει να το πει και χαίρομαι ότι κάποιος το είπε βεβαίως μου λέτε τώρα δεν είναι ένας υπεύθυνο, αλλά αυτός που φέρει την πολιτική ευθύνη έχει και τον πολιτικό συντονισμό Πιστεύω λοιπόν ότι θα μπορέσει η κυρία Άστον στο τέλος να προβεί στο συντονισμό. Είναι νέα βέβαια, είναι βαρύ το έργο και είναι σαφές ότι θα πρέπει να, γίνει, να είναι η επικεφαλής της ομάδος Ρέλεξ και θα πρέπει σε κάποιο επίπεδο όλα αυτά να ε, αποτυπωθούν και εις ε, την πραγματικότητα της χορηγήσεως βοηθείας δεν μπορεί όμως όλα να τα κάνει μόνη της. Χρειάζεται καλές υπηρεσίες οποίες έχουμε και ενδιαμέσους επιτρόπους οι οποίοι θα μπορούν να λειτουργούν κάτω από τη δική της συντονιστική δράση κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά διότι δεν μπορεί ένα άτομο μόνο του να τα κάνει όλα συνάδελφοι, θα σας καλούσα να είστε σύντομοι και στις ερωτήσεις και στις απαντήσεις. Γιατί θα ήθελα να, να ε, δοθεί δυνατότητα σε όλους ε, να μιλήσουν. Αυτό είναι το σωστό. Κύριε Γκρέσ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα κανονικά θα έπρεπε να έχω 30 λεπτά για την ομάδα μου και με βάση αυτά που είπε ο κύριος Χατζημαρκάκης. Θα μας λείψετε. Να σας ευχηθώ ότι καλύτερο κυρία Επίτροπε είχαμε μια ε, μετριοπαθή φιλία. Υπήρχε όμως φιλία, φιλική σχέση στην Επιτροπή μας για τα θέματα εξωτερικής ε, ε, δράσης. Πολύ συχνά είδαμε ότι τίνατε ευήκον ους και αυτό θέλουμε να το συνεχίσουμε. Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο πακέτο, μας έχετε στο πλευρό σας, αλλά θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί γιατί δεν ξέρουμε με την εξωτερική αυτή υπηρεσία ε, τι μας περιμένει. Σε ό,τι αφορά την ε, μελλοντική αυτή εξωτερική υπηρεσία, χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες. Είδα το παράδειγμα 10 του καταστατικού. Σε ό,τι αφορά το καθεστώς των υπαλλήλων σε τρίτες χώρες, θέλω να κάνω λοιπόν κάποιες ερωτήσεις προς τις υπηρεσίες που αφορούν βεβαίως νούμερα, μέχρι τούδε επιδόσεις ε, και θα ήθελα να μου απαντηθούν για να μην ε, ζητήσω απάντηση ε, τώρα. Παρακαλώ να λάβουμε όλοι απαντήσεις σε ερωτήσεις που υπάρχουν ήδη. Τώρα, στην επιθεώρηση των αντιπρόσωπιών αναφέρεται ότι η κοινοτική είναι ε, απόντες στο 40% του χρόνου. Έκανα μια γραπτή ερώτηση σχετικά που δεν απαντήθηκε από την Κομισιόν και παρακαλώ τώρα να προβληματιστείτε λίγο για να δείτε τι είναι αυτή η τεράστια χρόνια απουσίας γιατί ε, ούτε μετεκπαίδευση, ούτε άδειε, ε, ούτε τίποτε άλλο, ε, υπηρεσιακά ταξίδια κλπ. υπολογίζονται εδώ. Ε, είναι άλλος χρόνος. Επίσης δεν ήξερα ότι 5.000 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε αντιπροσωπείες μαζί με τους ε, επιτοπίους Πόσοι λοιπόν σχεδιάζονται να είναι στην εξωτερική υπηρεσία, δηλαδή πόσους πρέπει να υπολογίζουμε. Καλό θα ήταν επίσης να ξέρουμε σιγά σιγά το θέμα των αποστολών ασφαλείας ε, αν ε, περιλαμβάνονται στον ε, προϋπολογισμό, τι δομές θα έχουν, αν θα, ε, πώς θα, ποια θα είναι η διαχείριση, θα διαχειρίζεται η Κομισιόν. Είναι σημαντικό αυτό και για τα ε, δικαιώματα ε, ελέγχου και διαχείρισης. Επίσης ο τομέας ρέλεξε Πώς θα περάσει στην εξωτερική υπηρεσία, γιατί μέχρι τώρα το καταστατικό δεν βλέπει κάτι τέτοιο. Ε, αναφέρεται στην εθελοντική δράση. Δηλαδή, ε, οι κύριοι που σε συνοδεύουν θα είναι υποχρεωμένοι, δεν θα είναι πλέον μια εθελοντική δραστηριότητα. Ήρθε η ώρα να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Δεν ξέρω, με την περασμένη Παρασκευή στην Κορεπέρα έγινε μια συζήτηση σχετικά με τη νέα εξωτερική υπηρεσία. Όλοι ξέρουν περισσότερα πράγματα από εμά. Και νομίζω ότι αυτό ε, στα πλαίσια της περαιτέρω διαδικασίας ε, της Κομισιόν δεν είναι δίκαιο. Ε, αξιότιμη κυρία Γκρέσλε, καταρχήν ευχαριστώ για αυτά που μου είπατε, ότι θα σας λείψω. Τώρα για την εξωτερική υπηρεσία, ε, εγώ είμαι η προκάτοχος και για το, τώρα μιλάμε για το 2008. Πρέπει να πω ότι για την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων πολλά θέματα δεν έχουν ακόμη απαντηθεί και διευκρινιστεί και κάποια στιγμή θα πρέπει να ε, δεχτούμε ότι η Lady Άστον δεν έχει ακόμα γίνει επίσημα ε, δεκτή, δεν έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο ακόμη, όπως και οι άλλοι επίτροποι. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, οπότε δώστε της λίγο χρόνο. Γενικά θα ήθελα να πω αυτό που γνωρίζω προσωπικά και ε, έχω και άποψη για να το πω στα αγγλικά το πρώτο. Καταρχήν, νομίζω ότι η ανάγκη και οι προκλήσεις ε, ε, τώρα με αυτή τη στρατηγική μηδενική ανάπτυξη του προσωπικού που υπάρχει εδώ και καιρό και εγκρίθηκε από την Κομισιό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη για όλους. Σε αυτό το πλαίσιο αριθμός μέτρων ελήφθη για τη βελτιστοποίηση της πολιτικής ανθρωπίνων πόρων ώστε να γίνει πιο ευέλικτη κυρίως με την κατάρτιση. Όμως παρόλα αυτά και αυτό είναι προσωπική άποψη οι υπηρεσίες της Κομισιόν και ειδικότερα η Europe Aid αντιμετωπίζουν μια κατάσταση όπου καλούνται να εφαρμόζουν πολύ περισσότερη αναπτυξιακή βοήθεια σε αιτήσια βάση χωρίς να μπορούν να αυξάνουν ανάλογα το προσωπικό τους. Εγώ προσπάθησα όσο μπορούσα να υπερασπιστώ το προσωπικό. Βεβαίως υπάρχει ο Επίτροπος για τον Προϋπολογισμό, υπάρχει συνολικός προϋπολογισμός. Το Συμβούλιο μας ζητεί να μην δίνουμε περισσότερα, να μην αυξήσουμε τις δαπάνες, αλλά από την άλλη πλευρά εδώ καλούμεθα να είμαστε όλο και πιο ε, συγκεκριμένοι να βελτιώνουμε τη βοήθεια συνεχώς, ενώ από την άλλη πλευρά δεν αυξάνεται το προσωπικό, ούτως ώστε να παρέχεται με πιο σωστό τρόπο η βοήθεια. Γι' αυτό στο Europaid ο λόγος για το προσωπικό για κάθε 10 εκατομμύρια ευρώ μειώθηκε από το 2004, όταν άρχισε η δική μου η όπου είχαμε 4,8 ανθρω... ε, ανθρώπους ετησίως και τώρα το ποσοστό είναι 3,8 τέλος του 2009 και πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας που βεβαίως απενεργοποιεί αν θέλετε το προσωπικό που καλείται πολλές φορές να κάνει όλο και πιο δυσχερείς ε, δραστηριότητες στις ε, ε, ευάλωτες χώρες, στις δύσκολες χώρες και γι' αυτό αρνούνται και να πάνε. Γι' αυτό μεταξύ άλλων έχουμε μόνο 26% ποσοστό κενών θέσεων, ιδιαίτερα στις λεγόμενες ευάλωτες χώρες. Υπάρχει και ένας άλλος παράγον που είναι σημαντικός. Στις κεντρικές υπηρεσίες για τους συμβάση υπάρχει τριετή σύμβαση. Καταρτίζονται οι άνθρωποι κανονικά, ξέρουν τη δουλειά τους και μετά βγαίνουν να πάνε να την κάνουν. Είναι πάλι πολιτική μου άποψη ότι αυτή δεν είναι ε, σωστή στρατηγική. Δεν μπορούσα να το αλλάξω αυτό, αλλά αν υπήρχε δυνατότητα να αλλάξει θα ήταν καλό. Ε, ενώ ε, ε, στις αντιπροσωπείες μπορούν πάλι επισυμβάσεις να παραμείνουν. Και πάλι είχαμε ένα ποσοστό κενών θέσεων. Αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα, για το μέλλον, όπως σας είπα, όλες αυτές οι καινούργιες δομές θα πρέπει να αποφασιστούν. Η Lady Ashton, ως είπατε εκπρόσωπο, καλείται όπω γνωρίζετε να υποβάλει πακέτο προτάσεων στο Συμβούλιο σε στενή προφανώς συνεργασία με το Κοινοβούλιο τον Απρίλιο. Οπότε υπάρχει μια ομαδική εργασία, αλλά πολλά πράγματα δεν έχουν ξεκαθαριστεί ακόμη. Είπε σαφώ στην ακρόασή τη, αυτό και αυτό είναι βέβαιο, ότι όντως η υπηρεσία εξωτερικών δράσεων θα είναι το ίδιο υπόλογη όπως ήταν και το έργο της Κομισιόν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, σύμφωνα με τη συνθήκη. Πώς θα γίνει στην πράξη αυτό, δεν το γνωρίζω ακόμη. Αυτή τη στιγμή ο διατάκτης είναι η ίδια η Κομισιόν, η οποία Κομισιόν αφεαυτής αναθέτει ε, η εντέλει στο Γενικό Διευθυντή το διατάκτη, ο οποίος Γενικός Διευθυντής μπορεί μετά να ε, ε, δώσει εντολή στην αντιπροσωπεία. Αλλά ακόμη οι δεν είναι σαφείς, δεν έχουν αποφασιστεί και δεν είμαι πια επίτροπος για τις εξωτερικές δράσεις, δεν ήμουν στην Κορεπέρ και δεν έχω έκθεση, δεν μου στέλνονται οι εκθέσεις και δεν ξέρω τι είπαν εκεί αλλά είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους σας πάρα πολύ και συμφωνώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και να υπάρχει και προσωπικό ασφαλείας. Ε, γύρισα από την Κεντρική Αμερική, πήγα στην Γουατεμάλα, πριν από λίγο στην Κοσταρίκα και στο Ελσαλβαντόρ και η Γουατεμάλα ειδικότερα είναι μια χώρα ε, όπου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ασφάλειας. Εκεί ε, λαμβάνουν χώρα ή περισσότερες βιοπραγίες στον κόσμο, δολοφονίες κλπ. Οπότε βεβαίως αν πάτε εκεί χρειάζεστε ασφάλεια. Το προσωπικό η πάλι χρειάζονται ασφάλεια. Εκ λοιπόν σήμερα μπορώ να πω ότι αν θέλουμε να κάνουμε καλή δουλειά θα πρέπει να έχουμε ε, σωστό επίπεδο ασφάλειας και πάντοτε νιώθω ε, υπόλογη για την ασφάλεια των δικών μου. Εις ό,τι αφορά την ε, βία ε, χαίρομαι διότι συνέβησαν ελάχιστα πράγματα. Όμως υπήρξαν περιστατικά και πάντοτε μπορείτε να βελτιώσετε το επίπεδο ασφαλείας και το μηχανισμό ασφαλείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε 10 λεπτά για 5 αιτήσει, οπότε παρακαλώ οι ερωτήσει να είναι πάρα πολύ γρήγορε και δίνει το λόγο στην κυρία Γιάλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Φερέρο Βάλτνερ και να της ευχηθώ κάθε τι το καλύτερο στη συνέχεια της αδειοδρομίας της και ελπίζω ότι θα μπορέσει να, να συνεχίσει το επικοδομητικό έργο που έχει κάνει μέχρι στιγμής. Αφού μιλάμε λοιπόν για την εργασία της ΡΕΛΕΞ θα ήθελα να χαιρετήσω εδώ την Πιλάρ Χουάρες Ντοράλ η οποία είναι η υπεύθυνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ΑΙΤ και η οποία υπήρξε θύμα του σεισμού ε, πρέπει να χαιρετήσουμε το έργο της και συγχρόνως να αναφερθούμε στο λαό της Θα ήθελα λοιπόν παρακαλώ αυτό να γραφεί στα πρακτικά, διότι πολλές φορές για λόγους δημοσιονομικούς υπάρχουν ομάδες οι οποίες δεν είναι ασφαλείς. Ερχόμενοι τώρα στο έτος 2008, θα ήθελα κυρία Πρόεδρε να κάνω ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένα θέματα όσον αφορά τις σχέσεις με ε, τα ε, Ηνωμένα Έθνη. Ε, θίξατε ένα μέρος, αλλά θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται με τους ελέγχους, διότι το ελεγκτικό συνέδριο και πολύ σωστά λυπάται διότι δεν έχει πρόσβαση στην τεκμηρίωση, στα έγγραφα επειδή είμαι εισηγήτρια, ξέρω ότι τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίσαμε για το γραφείο του Κωσυφοπεδίου. Ξέρω ότι εσείς φεύγετε, αλλά χάρη στην πείρα σας μπορείτε να δώσετε συμβουλές. Τι να γίνεται κατά τρόπον ώστε η έλεγχη αυτή να είναι λιγότερο αδιαφανής και να μην αμφισβητεί κανείς την ε, αναγκαία συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό ήταν το πρώτο θέμα. Δεύτερον, όσον αφορά τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ξέρετε ότι υπάρχει το προσωπικό της Επιτροπής, οι συμβασιούχοι, Υπάρχουν όμως και άλλες οργανώσεις που είναι μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται επί τόπου. Αυτή τη στιγμή λόγω των προβλημάτων που έθιξε ο εισηγητής αμφισβητούμε την αποτελεσματικότητα αυτών των οργανώσεων. Υπάρχει μάλιστα και μία έκθεση που είχε παρουσιάσει ο κύριος Ντεγκούχτ ο οποίος έλεγε ότι θα πρέπει να μειώσουμε τους κινδύνους. Σας παρακαλώ να είστε σύντομοι γιατί διαφορετικά δεν θα προλάβουν οι άλλοι συνάδελφοι να παρέμβουν. Πρέπει να δώσω το λόγο σε τρεις παρεμβαίνοντες. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ποιο είναι το κίνδυνος ε, ε, για ε, αυτήν την παρέμβαση. Ευχαριστώ. Λυπούμε ιδιαιτέρως για την Ισπανίδα υπεύθυνο εις την ΑΙΤ Τα συλληπιτήριά μας προς την οικογένειά της θα μας λείψει αλλά αλλά όσον αφορά τα Ηνωμένα Εθνή, καταρχήν θα ήθελα να αναφερθώ στην πρόσβαση. Δηλαδή, πολλές φορές διαπιστώσαμε ότι ήταν δύσκολο να έχουμε πρόσβαση. Δηλαδή, δεν υπήρχαν πολλά γραφεία τα οποία δεν αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικό είναι το θέμα. Έχουμε συνεργαστεί με τα Ηνωμένα Έθνη. Ε, με τα Ηνωμένα Έθνη. Έχω εγώ προσωπικά συνεργαστεί με τον Γενικό Γραμματέα και ο Διευθυντής μου έχει συνεργαστεί με άλλα κλιμάκια θα έπρεπε λοιπόν το ελεγκτικό συνέδριο να έχει πρόσβαση στα στοιχεία, στα δικαιολογητικά. Διότι ακόμη και είναι δύσκολο όταν εμείς παρεμβαίνουμε πάντοτε βοήθησε ιδίως στο Μπαγκλαντές. Οι έλεγχοι μέχρι τώρα έχουν πάει πολύ καλά και ελπίζουμε να καταλάβουν διότι τους είπαμε σαφέστατα. Αν δεν λειτουργήσει αυτό σωστά τότε και εμείς θα χρειαστεί να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Τώρα, για τους κινδύνους και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ξέρετε ότι το σημαντικότερο είναι η απόφαση για την παροχή κάποιας επιχορήγησης να στηρίζεται σε πάρα πολύ καλή διαδικασία επιλογής με βάση τις προτάσεις που θα ζητηθούν. Και η αξιολόγηση γίνεται μετά από μια ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγηση, των οποίων τα μέλη είναι επαγγελματίε, ειδικοί. Η απόφαση λαμβάνεται λοιπόν πάνω στη βάση της οικονομικής και τεχνικής αξιολόγησης της πρότασης που υπευλήθη χωρίς καμία πολιτική επιρροή από την πλευρά μας. Έτσι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Έτσι ε, λειτουργήσε το σύστημα και λειτουργήσε καλά. Ευχαριστώ κύριο Σεσόντεργα. Σα παρακαλώ πολύ γρήγορα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο για τις προσπάθειές της. Να κάνω μία ερώτηση όσον αφορά τα κονδύλια για την Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004 στο διάστημα 2004-2012 Ε, ακούγεται τώρα γιατί υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα. Μάλιστα, ωραία, αφού ακούτε, συνεχίζει ο μιλητή. Ήθελα λοιπόν και εγώ να ευχαριστήσω την Επίτροπο και να κάνω μία ερώτηση όσον αφορά τα κονδύλια για την Τουρκία. Επίτροπε, στη γραπτή μας απάντηση μιλήσατε για για ένα σημαντικό ποσό ε, και φαίνεται ότι μέσα από την απάντησή σας ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει η ικανότητα διαχείρισης, ε, ορθής διαχείρισης των χρημάτων αυτών στην Τουρκία. Αλλά πρέπει να σας πω ότι το, το Σουηδικό Ραδιόφωνο έκανε μία, ε, μία έρευνα και φάνηκε ότι ε, το πρόβλημα έχει να κάνει με τη χρησιμοποίηση της βοήθειας και με απάτες. Δηλαδή, με δύο λόγια, τα κονδύλια αποτελούν αντικείμενο πολιτικής, ε, ε, ε πολιτικής εκμετάλλευσης. Δίδονται δηλαδή εκεί όπου ελέγχονται από το Ισλαμικό κόμμα τα χρήματα. Ενώ οι υπόλοιποι δεν παίρνουν τίποτα. Θέλω λοιπόν να σας ζητήσω να σχολιάσετε το ζήτημα αυτό. Και κάτι άλλο. Φαίνεται όμως ότι φαίνεται ότι η επίτροπο δεν ε, είναι ικανοποιημένη από τον ορισμό του σφάλματος. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω ποια είναι η θέση του Συμβουλίου σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Σα παρακαλώ, δεν είμαι υπεύθυνη εγώ για το θέμα αυτό. Ε, ο επίτροπο Ρεν είναι ε, υπεύθυνο για τη διεύρυνση, άρα και για τα κονδύλια τα οποία διοχετεύονται στην χώρα αυτή. Σα ζητώ συγγνώμη, δεν είμαι υπεύθυνη εγώ, λέει η κυρία... Αναφέρει η κυρία Επίτροπο Αμα κοιτάξτε στην απάντηση που, εδώ, που δώσατε, στη γραπτή απάντηση, αναφέρεστε στο ζήτημα αυτό. Οπότε δίνετε ήδη μια απάντηση, γι' αυτό εγώ έκανα τη διευκρίνηση. Επόμενη ερώτηση, κύριε Ντράσνερ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε, είπατε ότι καταβάλλετε κάθε προσπάθεια Τι κάνετε το καλύτερο που μπορούσατε και ελπίζω να είναι να ισχύει. Αλλά φαίνεται όμως και με βάση τις γραπτές απαντήσεις δεν αρκούν όλα αυτά. Στην ερώτηση 2 είπατε και μας παραπέμπετε στην ε, έκθεση, στον ελέγχο, στην έκθεση ελέγχου 22 πρώτου 2009 όσον αφορά τη συνεργασία με το Ηνωμένα Έθνη και λέτε ότι δηλαδή τι λέτε εδώ ότι από 2009 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει άλλος έλεγχος και η αρχική έκθεση ήταν τον Ιούλιο του 2006 και τελικά είχαμε την έκθεση το 2009. Πέρασαν λοιπόν τρία χρόνια. Στο σημείο 3 αναφέρεστε στη δημιουργία μιας μονάδας που, που είναι ενεφερεμένη στους ε, ελέγχους ex Γιατί τώρα ε, αυτό έγινε το 2007 και όχι πριν. Και επίσης, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, στο 4 αναφέρεστε στο CRIST, στο Common Relics Information System, στο κοινό πληροφοριακό σύστημα ε, και στις κριτικές του ελεκτικού συνεδρίου. Το ε, όμως ε, αυτό δημιουργήθηκε μετά από την έκθεση άμυς έλεγχος για τα πληροφοριακά συστήματα και συστήματα διαχείρισης του συνεδρίου. Ε, τώρα, τι λέτε. Εσείς λέτε εδώ ότι, πρόκειται, ότι αυτό, αυτός ο οργανισμός έγινε πριν 1,5 χρόνο, μα έχει ιστορία 7 ετών. Και ρωτώ, τι γίνεται με το προσωπικό και τι ανάγκες υπάρχουν. Και αναφέρομαι σε αυτά τα οποία είπατε και πριν από λίγο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Όσον αφορά το πρώτο σημείο, να σας πω με σαφήνεια. Ο έλεγχος για την ε, υλοποίηση ναι, η, η τελική ε, πρόταση έγινε στις 28 Ιουλίου. Είχαμε και την τελική έκθεση ελέγχου και τελικά φτάνουμε στις 22 Ιανουαρίου του 2009. Από τις αρχικές 10 υποδείξεις δεχτήκαμε τις 8, η ΕΤΚΟ, εμείς και η ΕΚΟ. Και υπήρξαν τρεις συστάσεις ανοιχτές όσον αφορά το σχεδιασμό και το αποτέλεσμα των επαληθεύσεων και για την ενοποίηση δηλαδή, η ε, ε, ε, παγιοποίηση των προσπαθειών μας και στις δύο προσπάθειες και ε, οι υπόλοιποι δύο θεώρησαν ότι μπορούν να κλείσουν και αυτές τις στάσεις. Όσον αφορά τη συνολική αξιολόγηση ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και εταίρων, ε, αυτό που είπαμε ήταν να γίνονται περαιτέρω εκθέσεις για τις επιμέρους ικανότητες και να δημοσιεύονται τα αποτελέσματα για να αποτελούν τη βάση για τις σωστές αποφάσεις και βεβαίως μετά από αξιολόγηση των εταίρων των ΗΠΑ π.χ. στον Παγκλατές και στην Ιγυρία και μετά από διάφορες αναλύσεις φάνηκε ότι ε, η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ θεωρεί ότι ε, εφαρμόστηκαν οι συστάσει. Και όσον αφορά την ερώτηση, το ζήτημα για τις διαβεβαιώσεις από τα Ηνωμένα Έθνη και τις διασφαλίσεις, μπορώ να σας πω ότι έχουμε το σύστημα του τέταρτου πυλώνα, ε, του τεσσάρων πυλώνων, που, ε, όσον αφορά τα διάφορα στάδια και έχουμε δώσει οδηγίε στι αντιπροσωπείε. Με δύο λόγια θέλω να πω ότι βελτιώσαμε ιδιαίτερα το σύστημα και ελπίζω, όπω σα είπα, ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ε, Σα έδωσα όλα τα πολιτικά επιχειρήματα τα οποία ε, ε, ε συνηγορούν προ την κατεύθυνση αυτή και νομίζω ότι εδώ πραγματικά δεν μπορούμε να, ε, να πούμε ότι δεν θα εργαζόμαστε πλέον με τα Ηνωμένα Έθνη. Δεύτερον, για τον ειδικό ε, έλεγχο ex post που δημιουργήθηκε το 2007 στη Γενική Διεύθυνση Ρέλεξ ήταν άμεσο αποτέλεσμα του follow-up των διαφόρων ελέγχων. Άρα λοιπόν Λοιπόν, ε, και εδώ η Επιτροπή εφάρμοζε το πρόγραμμα δράσης. Εργαστήκαμε λοιπόν με βάση το συγκεκριμένο έλεγχο και φαίνεται η εργασία αυτή τώρα είναι ικανοποιητική και, και συμφωνεί ε, ότι είναι ικανοποιητική και το συνέδριο. Εργαζόμαστε με πολύ λίγα χρήματα, μην το ξεχνάτε. Ε, στο μεταξύ, τότε εργαζόμαστε με πολύ λίγα χρήματα σε επίπεδο ΚΕΠΑ. Τώρα λοιπόν έχουν αυξηθεί τα πράγματα. Και όσον αφορά το ΚΡΙΣ, και την ποιότητα των δεδομένων σε αυτό το Common Relics Information System, το CRIS, η βασική βελτίωση πρέπει να αφορά τα ε, επιχειρησιακά ε, δεδομένα. Η βελτίωση των δεδομένων αποτελεί ε, κύριο στοιχείο της προσοχής μας, και αποτελούσε αυτή εξ αρχή. Αλλά καταλαβαίνετε, απαιτείται κάποιο χρόνο. Μέχρι τελικά να καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου ε, έχουμε συστηματοποιήσει τι προσπάθειέ μα. Για παράδειγμα, αυτό το οποίο κάναμε και προσέξαμε ιδιαίτερα τι λεπτομέρειε, είχαμε πλαίσιο για ποιότητα δεδομένων, αυτό το φτιάξαμε, διαδικασίε για διαχείριση των δεδομένων ε, και εδώ προβλέπονται και έλεγχοι για την ποιότητα των στοιχείων, ε, για το ξεκαθάρισμα των στοιχείων, διαχείριση των δεδομένων και εδώ λοιπόν πρέπει να πω ότι βελτιώσαμε το σύστημά μας σημαντικά. Ευχαριστώ. Επόμενο ομιλητή, ο κύριο Οντή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ με τη σειρά μου. Θα ήθελα, ε, κυρία Βάλτνερ, να σας πω ότι ε, πολλοί είμαστε αυτοί που ε, ε, ε πιστεύουμε ότι θα μας λείψετε, θα μας λείψει η δέσμευση με την οποία ε, ε, ε, ασκήσατε τα καθήκοντά σας. Θα μας λείψει η κομψότητά σας, ο τρόπος με τον οποίο ασκούσατε ε, τα, τα καθήκοντά σας. Πραγματικά σας βλέπουμε στην τηλεόραση και αισθανόμασταν υπερηφάνεια που ήμασταν Ευρωπαίοι. επειδή είχα πολλές ερωτήσεις, αλλά είπε πρώτα πριν να βιαστούμε, να, σας, ρωτήσω λοιπόν για τα ασφάλματα και έχετε δίκιο που αρχίσατε αυτή την προβληματική με το συνέδριο. η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή. Επίτροπε, Είμαστε πολλοί αυτοί που περιμένουμε την πολιτική σας διαθήκη κατά κάποιο τρόπο. Και ε, στις επόμενες ε, ε, απαλλαγές πάντα το ερώτημα προς την Επιτροπή ήταν σαφές. Δεν ήρθε η ώρα να δημιουργηθεί ένα κοινοτικό μέσο, κοινοτικό όργανο για την εξωτερική δράση. Στην περασμένη απαλλαγή δεν απάντησε η Επιτροπή. Σε ρωτώ, δεν πιστεύετε ότι απαιτείται ένα κοινοτικό όργανο για να συγκεντρώνει όλα αυτά τα οποία γίνονται από την Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, από το διακυβερνητικό επίπεδο, το κοινοτικό επίπεδο. Εμείς λοιπόν, εμείς που είμαστε ευρωβουλευτές, τα έχουμε χαμένα. Καταλαβαίνετε τι αισθάνεται ο απλός πολίτη. Τι άποψη έχετε για το συγκεκριμένο θέμα. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα Καταρχήν για το, τη φιλοφρόνηση αυτή που μου απευθύνατε Όντως θα μου λείψει ότι δεν θα είμαι πλέον εδώ. Ε, αλλά σχετικά με την ερώτησή σας πιστεύω ότι πρόκειται για ένα πολύ περίπλοκο εργαλείο και για να μπορέσουμε να καταρτήσουμε ένα ενιαίο εργαλείο θα έπρεπε να προβούμε σε μία πολύ εκ των ε, ε, βαθέων ανάλυση των δυνητικών επιπτώσεων. Δεν λέω ούτε ναι ούτε όχι, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα μπορούμε να το ζητήσουμε από όλους εμπειρογνώμους από τον εαυτό μας, από το ελεγκτικό συνέδριο, ίσως θα πρέπει να προβεί σε μία ανάλυση και να δούμε πού θα καταλήξει, υπέρ και κατά. Νομίζω ότι αυτή είναι η ειλικρινής απάντηση που μπορώ να σας δώσω. Όσον αφορά το θέμα, είναι όντως ε, σημαντικό, χρειαζόμαστε περισσότερη συνεκτικότητα, περισσότερη εναρμόνιση, αλλά δεν ξέρω ε, αν μετά από την συνέχεια οι λεπτομέρειες ίσως ε, δεν θα καλύπτονταν. Ευχαριστούμε. Σα ευχαριστώ και εγώ για την ακρόαση αυτή και να δώσω αμέσω το λόγο στον κύριο Σάρμα, στον εκπρόσωπο του συνεδρίου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού, έχω κληθεί εδώ για να σας παρουσιάσω τις παρατηρήσεις του ελεκτικού συνεδρίου που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 11 σχετικά με τις διοικητικές δαπάνες ε, στο, στην ετήσια έκθεση. Όσον αφορά το κεφάλαιο 11 θα βρείτε τέσσερις κατηγορίες πληροφοριών. Καταρχήν όσον αφορά τις συναλλαγές δεύτερον όσον αφορά τα μέσα εσωτερικού ελέγχου δεύτερον σχετικά με τις, τους ειδικούς ελέγχους που έκανε το ελεγκτικό συνέδριο και ε, τη συνέχεια που δόθηκε στις προηγούμενες παρατηρήσεις που είχε διατυπώσει το ελεγκτικό συνέδριο όσον αφορά τις συναλλαγές ε, το συνέδριο ήλεγξε το 2008 ο, πέραν ε, των 500 συναλλαγών και τα αποτελέσματα αυτής, αυτών των ε, ελέγχων ήταν ότι ε, δεν υπήρξαν ε, σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή όσον αφορά τις συναλλαγές που ελέγχθηκαν δεν είχαμε σοβαρά προβλήματα. Όσον αφορά τους εσωτερικούς ελέγχους ε, το ελεγκτικό συνέδριο δεν διαπίστωσε ε, σημαντικές ελλείψεις. Τρίτον, ελέγξαμε μία σειρά από συγκεκριμένα θέματα και θα δείτε το αντικείμενο του ελέγχου μας στο κεφάλαιο 11 στο κάτω μέρος της σελίδας όπου αναφερόμαστε στους ελέγχους διαφόρων θεσμικών οργάνων και όπου λέμε ότι οι ε, διαπιστώσεις του ελεγκτικού συνεδρίου έγιναν αποδεκτές από τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα και τώρα παρακολουθούμε πώς οι παρατηρήσεις παρατηρήσεις αυτές στη συνέχεια εφαρμόστηκαν από τις διάφορες εμπλεκόμενες από τα διάφορα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα. Και τέλος, όσον αφορά αυτές τις παρατηρήσεις μας, το τελευταίο σχόλιο είναι ότι διαπιστώνουμε μία πρόοδο στα πιο σημαντικά θέματα και το συμπέρασμα συνολικά, το οποίο μπορώ να αναφέρω όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες, είναι ότι ότι η γενική αντιμετώπιση του ελεγκτικού συνεδρίου είναι ε, θετική. Πρέπει να τονίσω επίσης από πλευράς μεθοδολογικής κάτι βασικό κατά τη γνώμη μου, δηλαδή ότι το συνέδριο εκδίδει ένα συνολικό συμπέρασμα για όλα τα θεσμικά όργανα και όχι για ένα θεσμικό όργανο μετά το άλλο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε το λεκτικό συνέδριο. Να δώσω τώρα το λόγο στο Γενικό στη Γενική Γραμματέα της ε, Επιτροπής, την κυρία Κατεναντέη, την οποία ήθελα να ε, καλωσορίσω. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλό σας απόγευμα. Χαίρομαι που έρχομαι πάλι εδώ στην Επιτροπή σας. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας απόψε. Τώρα, στη μεταβατική περίοδο από τη μία Επιτροπή στην άλλη, εγώ αντιπροσωπεύω τη συνέχεια του συστήματος, υποθέτω, και είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνετε να πω δύο λόγια σχετικά με το τι κάναμε τον τελευταίο καιρό για να βελτιώσουμε διαχείριση και έλεγχο των οικονομικών της Κομισιόν που είναι η ευθύνη μας και η αρμοδιότητά μας. Είχα την ευκαιρία να πω ήδη παλιότερα και ελπίζω να σας πείσαμε. Χρησιμοποιούμε σημαντικούς πόρους για τη διαχείριση και διοίκηση που θεωρούμε πολύ σημαντική και νομίζω ότι υπάρχουν και αυτά αποτελέσματα. Η Κομισιόν με πολύ ομαλό τρόπο αντιμετώπισε ε, τα προβλήματα πρόσφατα και τα τελευταία χρόνια είχαμε σταθερούς πόρους για να δώσουμε καλά πολιτικά αποτελέσματα. Δεν είναι όλα τέλεια θα είμαστε οι πρώτοι που θα το αναγνωρίσουμε αυτό και θα επιδιώξουμε σε αιτήσια βάση και άλλες βελτιώσεις, γιατί παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας ακόμα η Κομισιόν δεν έχει λάβει χωρίς επιφυλάξεις ε, ε έκθεση αξιοπιστίας από το ελεγκτικό συνέδριο. Εσείς όμως θα παρακολουθείτε αυτά σε κανονική μακροπρόθεσμη βάση και γι' αυτό νομίζω ότι μπορείτε να δείτε τις προσπάθειες που κάνουμε για τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και είμαι βεβαία ότι με τον ίδιο πρόεδρο επικεφαλής η Νέα Κομισιόν θα ακολουθήσει την ίδια προσέγγιση με αποφασιστικότητα και, και ανανεωμένο σθένος. Μας ενθάρρυνουν οι τελευταίες οι εκθέσεις του ελεκτικού συνεδρίου που δείχνουν σαφώς την πρόοδο που έχει επιτελεστεί και τα θετικά αποτελέσματα των κοινών προσπαθειών μας στα διάφορα θεσμικά όργανα για να βελτιώσουμε τη διαχείριση των κονδύλιων. Θεωρώ ότι αυτό οφείλεται σε έναν αριθμό σημαντικών μέτρων που συζητήθηκαν με την Επιτροπή σας ε, κατά τη διάρκεια των ετών και που ε, υλοποιήθηκαν από την Κομισιόν. Αναφέρω ορισμένα από αυτά που σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και θα είμαι ευτυχής να επανέλθω και αργότερα σε αυτά τα θέματα. Καταρχήν πιστεύω ότι ε, χρόνο με το χρόνο βελτιώσαμε την κάλυψη και την ποιότητα της ε, έκθεσης σύνθεσης όπου αναλαμβάνει η Κομισιόν Πολιτική Ευθύνη για τη διαχείριση των κονδυλίων από τις υπηρεσίες της και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που βλέπουμε ότι το ελεγκτικό συνέδριο αναγνώρισε την συνεχή βελτίωση και την ποιότητα τη ετήσια έκθεση πεπραγμένων που υποβάλλεται από του γενικού διευθυντέ κάθε χρόνο ως ε, συνοδευτικά της Γενικής Έκθεσης. Επίσης εφαρμόσαμε το σχέδιο δράση του 2006 για ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου και νομίζω ότι είναι δυνατόν επί τη βάση αυτού του προγράμματος δράσης να καταδείξουμε ότι τώρα έχουμε πολύ πιο ισχυρό σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Επίσης ξέρω ότι η Επιτροπή παρακολούθησε εκ του σύνεγγης το πρόγραμμα δράση του 2008 της Κομισιόν για να ενισχύσουμε τον εποπτικό ρόλο για διαρθρωτικέ δράσεις της Κομισιόν. περισσότερες δράσεις έχουν ολοκληρωθεί τώρα, αλλά ακόμα συνεχίζονται οι εργασίε και η πρόθεσή μας είναι να υποβάλουμε νέα έκθεση ε, προόδου ε, στην αρχή μετά την ε, σύνθεση της Κομισιόν. Πρώτη τελευταία παρατήρηση, οι, οι ετήσιες δηλώσεις αξιοπιστίας και οι συνοπτικοί πίνακες και είναι σημαντικοί για την διαχείριση και με τον Επίτροπο ε, Κάλλας ε, κάναμε πολλά για να βελτιώσουμε τη διαφάνεια του συστήματος, ε, δίνοντας δεδομένα για τους δικαιούχους, για ποσά τα οποία διαχειρίζεται κεντρικά η Κομισιόν. Υπάρχει ένα πόρταλ στο website το οποίο συνδέει με τα εθνικά website, όπου όλα αυτά είναι διαθέσιμα. Ένα καινούριο τομέας που θα μας απασχολήσει φέτος είναι μια συνέχεια στην αντίληψη της Κομισιόν σχετικά με ανεκτήματα. Ε, ανοιχτούς κινδύνους φαλμάτων ε, το 2008 με βάση το 2008 και θα δούμε ποια θα είναι η σωστή ισορροπία μεταξύ κινδύνου και κόστους ελέγχου. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι προβληματικοί τομεί που ενδιαφέρουν την Επιτροπή σα. Καταρχήν, είμαστε αποφασισμένοι να βελτιώσουμε την κατάσταση στα διαθροτικά ταμεία. Ξέρω ότι οι Επίτροπη για την Ανάπτυξη σα ενημέρωσαν ε, σχετικά με το πώς επικεντρώνουμε τις δραστηριότητές μας σε τομείς με υψηλό ρίσκο ε, σφάλματος και πώς ενισχύουμε και το σύστημα ανάκτησης ε, χρεωστήτως καταβληθέντων. Η Νέα Κομισιόν οπωσδήποτε πολύ γρήγορα θα φροντίσει το θέμα της απλούστευσης της νομοθεσίας εκεί όπου πιστεύουμε ότι κάποιες αλλαγές θα μειώσουν το κόστος ελέγχου και τα σφάλματα στις συναλλαγές τις δημοσιονομικές οικονομικέ. Θέλουμε επίσης να κάνουμε προτάσεις για νέα απλούστευση των κανόνων επιλεξιμότητας ως μέρος της αναθεώρησης τριετούς ε, ε, του κανονισμού, του δημοσιονομικού κανονισμού και επίσης ε, δουλεύουμε πάνω σε ιδέες για μηχανισμούς παράδοσης πιο απλού, απλοποιημένους στα πλαίσια του ε, πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου. Όπως προείπα θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε ιδέες σε σχέση με το ανεκτό επίπεδο εσφάλματος και κίνδυνο σφάλματο, γιατί αυτό είναι σημαντικό για να έχουμε καλύτερη ισορροπία από το σήμερα μεταξύ δαπανών ελέγχου και ε, υψηλά επίπεδα ελέγχου σχετικά με ρίσκο για τον κοινωνικό προπολογισμό. Φέτος λοιπόν θα υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις για πολλές διαρθρωτικές πολιτικές και με χαρά θα συνεχίσουμε τη συζητήση μας με την Επιτροπή σας κύριε Πρόεδρε. Αυτά ήθελα να πω ως εισαγωγή στο θέμα, χωρίς να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες εκτός και αν το θελήσετε. Ευχαριστώ κύριος Λιμπεράσκη. το λόγο για τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Γενική Γραμματέα, Ας ξεκινήσουμε από αυτό που είπατε στην αρχή της ομιλίας σας για τη συνέχεια. Αναμφίβολα, η συνέχεια ε, αποτελεί πλεονέκτημα γιατί ε, αλλάζουν οι επίτροποι και αλλάζουν και φυλάκια. Χαίρομαι λοιπόν για αυτή τη συνέχεια. Τώρα, κώδικας διοντολογίας για τους ε, επιτρόπους. Οι υπηρεσίε τη Επιτροπή θα προτείνουν ένα νέο κώδικα δεοντολογία λαμβάνοντα υπόψη πτυχέ όπω έλλειψη ορισμού του όρου σύγκρουση συμφερόντων. Δηλαδή, σκέφτεστε να δώσετε συγκεκριμένο περιεχόμενο, ακριβέ περιεχόμενο στον όρο αυτό. Εάν δεν υπάρξει ε, πώς θα υπάρξει περιγραφή ε, μιας πορείας δράσης εάν υπάρξει σύγκρουση συμφερόντων. Μα τι θα μπει σύγκρουση συμφερόντων και αν προκύψει θα γίνει συνέχεια. Επίσης υπάρχει έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά το θέμα της αποδοχής δώρων. Φιλοξενίας ή κάποιου άλλου στοιχείου. Πώς θα διακρίνουμε τις περιπτώσεις. Επίσης, η Επιτροπή θα αναθεωρήσει, θα, θα δεχθεί, θα εγκρίνει το, αναθεωρημένο κώδικα δοντολογίας ε, μέχρι το τέλος του 2010. Πρόεδρε, μετά μου επιτρέψετε θα κάνω και κάποιες συμπληρωματικές ερωτήσεις. Thank you very much. Well, uh, Σας ευχαριστώ. Όπως ξέρετε, η Επιτροπή διαθέτει κώδικα δεδολογίας, ο οποίος αναθεωρήθηκε πριν από λίγα χρόνια και που εφαρμόζεται με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο. Όπω ξέρετε, στι πολιτικέ κατευθυντήριε γραμμέ για την επόμενη Επιτροπή, ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει στον κώδικα αυτό και μιλά βεβαίω για τη δυνατότητα αναθεώρηση υπό το φω τη εμπειρία. Ταυτόχρονα όμω, αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον είναι να δούμε τι ευκαιρίες θα υπάρξουν ε, για συζήτηση του κώδικα σε περισσότερο διοργανική και διαθεσμική βάση. Δεν μπορώ τώρα να σας πω εγώ πότε θα λάβουν χώρα όλα αυτά. Πάντως ε, εργαστήκαμε ιδιαίτερα ε, στο θέμα της διοντολογίας σε πέντε Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, κάναμε και, προχωρήσαμε σε έργο σύγκρισης. Φαίνεται λοιπόν ότι ήδη υπάρχει αυστηρός έλεγχος τη επιτροπής και αυτό μπορεί να αποδειχθεί μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχουμε ακολουθήσει και εφαρμόσει πολύ ψηλά πρότυπα διδολογία και ηθική. Σα παραπέμπω λοιπόν σε αυτά τα οποία είπε ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κατευθυντήριε Γραμμέ και να σα πω για άλλη μια φορά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την πρόθεση να αναθεωρήσει τον κώδικα υπό το φω τη εμπειρία μα, αλλά δεν μπορώ να σα πω πότε θα γίνει αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ναι, Κατάλαβα τι είπατε. Είπατε ότι υπάρχει ο κώδικα και την άλλη είπατε ότι θα αναφερθεί, παρόλο που δεν είπατε πότε. Τώρα, θα έχουμε μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο καταμερισμό των αρμοδιοτήτων και των χαρτοφυλακίων ανάμεσα στου επιτρόπου. Θα αναφερθώ σε αυτό. Είστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρξει καμία περίπτωση επικάλυψη αρμοδιοτήτων ή ότι δεν θα υπάρξει ποτέ σύγκρουση συμφερόντων. Για παράδειγμα, θα έχουμε επίτροπο υπεύθυνο για ε, την φοροδιαφυγή και ο ίδιος θα είναι υπεύθυνο και για τη φορολογία. Ε, πιστεύετε ότι αυτό ο συνδυασμό δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα? Απάντηση. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την κατανομή των χαρτοφυλακίων, νομίζω ότι ο πρόεδρος ε, ασχολήθηκε με διάφορες πτυχέ ε, και κύριο του μέλημα είναι να υπάρξει καταμερισμό ισορροπημένος καταμερισμός του φόρτου εργασίας ανάμεσα στου συναδέλφου. Και η, η, η, η γενική αντίδραση όταν ανακοίνωσε τα χαρτοφυλάκια είναι ότι πέτυχε το σκοπό του. Τώρα, στη σύγχρονη πολιτική, και αυτό το βλέπουμε ε, μέρα με τη μέρα, ε, τα, τα διάφορα ζητήματα αλληλοσυνδέονται. Και είναι πολύ δύσκολο να πει κανεί πού σταματούν τα σύνορα και τα όρια του ενό χαρτοφυλακίου και πού αρχίζουν τα, ε, και τα όρια του επομένου. Ακριβώ γι' αυτό η Επιτροπή λειτουργεί και δρά σαν σώμα. και γίνεται και προσπάθεια δράση με τη μορφή ομάδα επιτρόπων όσον αφορά σημαντικά ζητήματα στο παρελθόν ε, πρέπει να πούμε ότι υπήρξε πολύ επιτυχής ε, συνεργασία ε, αρκετών επιτρόπων σε ορισμένα ζητήματα, π.χ. ενέργεια και κλίμα, μετανάστευση κτλ. Άρα λοιπόν αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Εμένα, σε επαγγελματικό επίπεδο, δεν με απασχολεί το ζήτημα της πιθανής επικάλυψης χαρτοφυλακίων γιατί βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη αποφασιστικότητα από την ε, ε, καινούργια Επιτροπή για συνεργασία, ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από ό,τι στο παρελθόν. Και δεύτερον, δεν βλέπω να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων στα επιμέρους χαρτοφυλάκια για παράδειγμα, όταν έχουμε τον Επίτροπο υπεύθυνο για τους, για, τους δασμούς και τη φορολογία, ε, ο οποίος είναι και, και υπεύθυνο για την καταπολέμηση των, ε, της φοροδιαφυγής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Και ε, ε, μπορεί κανείς να είναι υπεύθυνο και για τα δύο αυτά χαρτοφυλάκια, χωρίς καμία σύγκρουση συμφερόντων και αρμοδιοτήτων. Ευχαριστώ. Κυρία Γενική Γραμματέα, μιλήσατε για την ανάγκη και τη βούληση εξοικονόμηση χρημάτων. Δηλαδή να είναι φθηνότερη η επιτροπή, λιγότερο δαπανηρή. Ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά τους εκτελεστικούς οργανισμούς. Οι εκτελεστικοί οργανισμοί γενικά τι ήταν επιτυχημένος θεσμός. Θα γίνουν κι άλλοι ή θα μειωθεί ο αριθμό τους και θα πείτε δεν θα φτιάξουμε άλλους. Ποια ήταν η αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά τα συμπληρωματικό κόστος και, ε, ε, ε, ποια ήταν η αποδοτικότητά τους. Απάντηση. Κοιτάξτε, δεν έχουμε και τόσου πολλού εκτελεστικού οργανισμού μέχρι στιγμή. Είναι σχετικά καινούργιο το φαινόμενο. Πάντω, όπω βλέπω εγώ το ζήτημα και η συνολική μα εντύπωση είναι ότι είναι αποτελεσματική και ε, αποδοτική. Νομίζω ότι η, η, ότι η εξέταση που έχει γίνει έχει δείξει ότι ε, με αυτόν τον τρόπο ε, η εφαρμογή ορισμένων ε, τομέων πολιτικής γίνεται με φθηνότερο τρόπο. λαμβάνοντα υπόψη ότι αυτά τα οποία αποτελούν αντικείμενο εξωτερική ανάθεση ε, ε, αποτελούν αντικείμενο τη περιγραφή. Πάντω νομίζω ότι η συνολική μα αξιολόγηση είναι ότι αποτελούν ένα χρήσιμο τρόπο διαχείριση τμήματων τη πολιτική και της δημοσιονομικής ατζέντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι θα έχουμε και άλλους ή ότι δεν θα έχουμε και άλλους. Γιατί τελικά αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να δούμε τι προκλήσει από υλοποίηση θα έχουμε στο μέλλον και κατά περίπτωση θα, θα βλέπουμε κατά πόσο πρέπει τα προγράμματα να αποτελούν το κείμενο διαχείριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή κατά πόσο είναι πιο αποτελεσματικό και από αυξικό του ωφέλου να γίνεται από του εκτελεστικού οργανισμού. Αν θέλετε λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν μέρο ε, των διαφόρων μέσων και εργαλείων που έχουμε για την ε, ε, εκτέλεση του ε, κοινοτικού προπολογισμού. Σε άλλε περιπτώσει είναι αποτελεσματική, σε άλλε περιπτώσει όχι. Άρα λοιπόν η απάντησή μου είναι ότι αυτό ε, εξετάζεται κατά περίπτωση και δεν υπάρχει ένα γενικό προσανατολισμό είτε υπέρ είτε κατά. Πάντω, μέχρι στιγμή η εμπειρία έχει δείξει ε, ότι ε, ε, και ο απολογισμό είναι θετικό. Ευχαριστώ. Κυρία Γενική Γραμματέα, θα ήθελα να απαντήσετε στις γραπτές μας ερωτήσεις, ε, διότι είπατε ότι από 40.000, 17.000 ε, προγράμματα την χάνουν διαχειρίσεως μέσω ευρωπαϊκής ε, ενισχύσεως. Μπορούμε να ξέρουμε πόσο διαχωρίζονται αυτά τα προγράμματα και, πόσο, και ποια ποια διαχείριση υπάρχει για κανένα από αυτά ή τουλάχιστον για την πλειοψηφία από αυτά. Ε, όσον αφορά ε, την πλειοψηφία των προγραμμάτων αυτών. Πρέπει να σας πω ότι δεν ξέρω. Λυπούμε γιατί ο κύριος Σουσόν που ήταν ε, εδώ πριν από πέντε λεπτά μπορούσε να έχει απαντήσει, αλλά θα κοιτάξω να σας απαντήσω γραπτός. Άλλη ερώτηση. Μπορώ αυτό που με ανησυχεί είναι οι εθνικές διαχειριστικές δηλώσεις τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη, όλα τα κράτη-μέλη, να παρουσιάσουν τις εθνικές δηλώσεις τους. Διότι ξέρουμε ότι οι δηλώσεις οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί δεν είναι ενοποιημένες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να καταρτήσει μία ενιαία μεθοδολογία η οποία θα συμβιβάζει τις δηλώσεις όλων των κρατών μελών. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με την ιδέα των εθνικών δηλώσεων αλλά δεν έχουμε πείσει ακόμη μέχρι στιγμής όλα τα κράτη-μέλη ότι πρέπει να τις χρησιμοποιήσουν και προς το παρόν είναι ε, εθελοντικές. Ε, δεν έχω υπόψη μου να, να έχει προσπαθήσει κανείς να τις εναρμονίσει. Προσπαθούμε να τις βελτιώσουμε όπου μπορούν να βελτιωθούν και να μπορέσουμε να τις αξιολογήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ε, το παράδειγμα που χρησιμοποιούμε προς τα άλλα κράτη-μέλη είναι καταρχήν να τους πούμε ότι είναι κάτι που είναι εφικτό, που είναι χρήσιμο και ε, είναι θέμα ε, χρηστής ε, διαχείρισης του κοινοτικού προπολογισμού. Προσπαθούμε λοιπόν να ε, προωθήσουμε την χρήση αυτών των δηλώσεων από όλα τα κράτη-μέλη χωρίς όμως να έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε ε, αυτή την μέθοδο. Και αν μου επιτρέπετε μία τελευταία ερώτηση, τουλάχιστον ε, ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε ε, μία, σε ένα θέμα συγκεκριμένο που είναι τον πυρηνικό σταθμό του Κοσλοντούι. Ε, ε, το, έθεσα την ερώτηση στον υποψήφιο επίτροπο Ταγιάννη, αλλά δεν μου απάντησε τόσο σαφώς. τι είναι οι προοπτικές χρηματοδοτήσεως μέχρι το 2035 και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις ευγενείς απαντήσεις που μας παρήχατε δεν έχω αντιληφθεί ακριβώς τι ζητάτε. Αυτό το οποίο ξέρω για το Κοσλοντούι είναι ότι ε, χρηματοδοτούμε την απενεργοποίησή του και έχουμε ε, συντονίσει ε, την, ε, ε, ε, την χρηματοδότηση αυτή με αυτήν άλλων παρεμφερών προγραμμάτων από ό,τι ξέρω όμως υπάρχει ένα πρόγραμμα μέχρι το 2013 δεν ξέρω αν εννοείται για το κόστος για να κλείσουν οι εγκαταστάσεις αυτές ή κάτι άλλο αν θέλετε μπορείτε να μου το διευκρινίσετε Ευχαριστώ τον κύριο Λιμπεράσκη και δίνω τώρα σε άλλους ευρωβουλευτές την κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ κυρία Γενική Γραμματέα. Χαίρομαι που είσαστε εδώ και έχω ερωτήσεις καταρχήν ε, στον μηχανισμό ε, ε, επαληθεύσεως με την Ρουμανία και τη Βουλγαρία όπου όπως λέτε και εσείς υπάρχουν πολλές παρατυπίες και μιλάτε για την καταπολέμηση της διαφθοράς ότι να, κοντεύουμε να συνηθίσουμε αυτό το θέμα αλλά θα έπρεπε να έχουμε πλέον αποτελέσματα διότι ζητήσαμε οι εκθέσεις να είναι εκθέσεις πρόοδου να μας λέγουν δηλαδή πού βρίσκεται η πρόοδος σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και την πρόθεση της δικαιοσύνης. Μπορείτε να μας δώσετε τέτοιες εκθέσεις πλέον προόδρου για μπορέσουμε να μετρήσουμε τα αποτελέσματα ε, και ε, γιατί η Όλαφ δεν ε, έχει συμμετάσχει στην εξαιρετική έκθεση για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Δεν ξέρω τι είναι η αλήθεια και τι όχι γιατί το Κοσλοντούι παραδείγματος χάρη δεν περιλαμβανόταν στην ειδική έκθεση για τη Βουλγαρία παρόλο που υπερβαίνει 56 εκατομμύρια. Ε, επίσης έχουμε ένα πρόβλημα με τον Γενικό Διευθυντή της ε, Όλαφ ε, ο οποίος έκανε ένα πραξικόπημα και δεν συμβουλεύθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αντικαταστήσει τον Γενικό Γραμματέα πράγμα το οποίο μας, δίνει, μας δημιουργεί προβλήματα με τον κανονισμό που ζητάει να είναι αμερόληπτος ο Γενικός Διευθυντής. Τώρα Άρα λοιπόν τι θα γίνει, θα πρέπει να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να υπάρξει ακύρωση ε, αυτής ε, της αναθέσεως. Ε, βέβαια ο κύριος Κάλλας μου λέει ότι δεν είναι πια υπεύθυνο, ο κύριος Εμέτα που θα είναι ο επόμενος μας λέει ότι δεν είναι ακόμη υπεύθυνο, άρα ποιος είναι υπεύθυνο. Μετά, εξωτερική υπηρεσία, το οποίο εσείς ηγείστε από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας σας εύχομαι από βάθους καρδίας καλή επιτυχία αλλά όλα μέχρι τώρα έχουν τύχει διαπραγματεύσεων και κλεισμένων των θεών των θυρών. Οπότε θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που τίθενται, πόσο πολύ μπορούν να αναπτυχθούν αυτές οι υπηρεσίες, αν υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου, πόσο ε, τελειώνει ο εσωτερικός κανονισμός, υπάρχουν ε, καταναγκαστικά μέτρα, προς το παρόν ξέρω μόνο για εθελοντικά και για μένα είναι πολύ βασικό να ξέρω ότι ο εντεταλμένος διατάκτης θα είναι, έχει αναλάβει τις εργασίες αυτές κατόπιν εντολής Ευρωπαϊκής Ενώσεως, διότι βλέπουμε αποτελέσματα. Πέστε μας πότε θα μπορέσετε να ενημερώσετε το Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε εμείς να βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο ενημέρωσης που είναι και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα μου πάρει λίγο χρόνο, αν μου επιτρέπετε, ελπίζω να μην έχουμε πρόβλημα για να απαντήσω. Τώρα, για τον μηχανισμό επαλήθευσης και συνεργασίας, όπως ξέρει πολύ καλά η κυρία Γκρέσλε, εδώ πρόκειται για πολύ δύσκολα θέματα σχετικά με την αλλαγή του νομικού και δικαστικού συστήματος και στα δύο κράτη-μέλη, που θα και, και τη θεσμοθέτηση ενό ολόκληρου συστήματος διαδικασιών ελέγχου. Δεν είναι ρεαλιστικό δηλαδή εδώ να περιμένουμε ταχεία πρόοδο. Αυτό που μπορούμε να έχουμε χάρη στην ε, μεγάλη συμμετοχή πολλών υπηρεσιών της Κομισιόν και με τις συνεργασίες ε, των ε, υπηρεσιών των κρατών μελών. Βλέπουμε κάποια πρόοδο. Δύο φορές το χρόνο υπάρχουν εκθέσεις, στέλνουμε στο Κοινοβούλιο. Τον Ιούλιο ε, κυρίως και μια ενδιάμεση την άνοιξη. Θα συνεχίσουμε, προτιθέμε να συνεχίσουμε αυτό το σύστημα. Πιστεύω ότι έχουμε καλή συνεργασία και με τα δύο κράτη-μέλη που προσπαθούν να αλλάξουν τα συστήματα που τα είχαν τόσο, τόσα χρόνια πριν. Από τη μία πλευρά θα πρέπει να υπάρχουν σωστοί νόμοι και οι κυβερνήσεις και στις δύο χώρες κάνουν προσπάθειες να αλλάξουν τον ποινικό κώδικα και να εξυγχρονίσουν το ε, δικαιικό σύστημα και να αλλάξουν και την ε, ε, δικαστική εξουσία με νέες προσλήψεις και να εφαρμόσουν βέβαια και τους νέους νόμους. Η Κομισιόν έδωσε έμφαση τα τεκμήρια της ε, υλοποίησης. Θέλουμε να υπάρχουν σωστές διαδικασίες, ώστε ο κάθε παραβάτης του νόμου θα προσάγεται στο δικαστήριο και αν βρεθεί ένοχος θα καταδικαστεί ανάλογα. Ένας από τους λόγους ε, που έχουμε ακόμα το μηχανισμό στις δύο χώρες είναι ότι ακόμα δεν είμαστε ικανοποιημένοι ότι ο βαθμός υλοποίησης είναι επαρκής και ότι η αλλαγή είναι μία αντιστρέψιμη. Πιστεύω ότι στις εκθέσεις ε, πρόοδου που δημοσίευσαμε νομίζω πέρσι το Σεπτέμβρη αποδεικνύεται η πρόοδος, αναφέρεται εκεί και ελπίζω ότι όταν ε, γίνει η ενημέρωση της έκθεσης το καλοκαίρι πάλι θα αναφερθεί περαιτέρω πρόοδος. Για να είμαστε δίκαιοι είναι μεγάλη κλίμακα του εξυγχρονισμού στις χώρες που θα πρέπει να γίνει σε πανεθνικό επίπεδο. Επίσης είναι πολύ δαπανηρές αυτές οι αλλαγές Δηλαδή θα πρέπει όλη η νομολογία να ε, περάσει σε σύστημα πληροφορικής για να είναι γνωστά, γνωστές οι αποφάσεις στις όλους τους δικαστές. Και βεβαίως ε, στη Ρουμανία που περνάει τώρα πολιτική λιτότητας δεν είναι εύκολο να ε, τηρηθούν οι ρυθμοί πρόοδου που θέλουν οι αρχές και εμείς. Πιστεύω πάντως ότι το βάθος της έκθεσης προόδου που, δημοσίευσε η Κομισιόν έχει βελτιωθεί πολύ τον τελευταίο 1,5 χρόνο, γιατί τώρα έχουμε σε μεγαλύτερο βάθος κατανόηση του συστήματος που και τώρα προσαρμοστήκαμε και στη συνεργασία μας με τις αρχές των δύο χωρών. Τώρα, για την Όλαφ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια περίπτωση κάποια κατάσταση ανησυχητική η οποία θα οδηγήσει σε απόφαση του δικαστηρίου. Είναι αρμοδιο... η ευθύνη της Κομισιόν να διασφαλίσει ότι η υπηρεσία θα συνεχιστεί όταν υπάρξει κάποιο τραγικό γεγονός όπως ε, θάνατος Γενικού Διευθυντού. Υπάρχουν οι αποφάσεις. Ο κύριος Μπρούνερ, ο Γενικός Διευθυντής, ήδη είχε ε, διορίσει κάποιον για να τον αντικαθιστά Κατά την απουσία του, η Κομισιόν ακολούθησε ε, αυστηρά τους κανόνες για τη συνέχεια της υπηρεσίας. Διαβουλευθήκαμε με τις νομικές υπηρεσίες που ε, διαβεβαίωσαν ότι η Κομισιόν σε αυτή την περίπτωση ακολούθησε τη σωστή διαδικασία, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτε το ανησυχητικό εδώ. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συνεχιζόμενη ε, λειτουργία και τη συνεχιζόμενη προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Τώρα, και ο, ο, και ο νέος επίτροπος είπαν ότι τώρα θα επιταχύνουμε τη δημοσίευση για την ε, κάλυψη της θέσης του νέου Γενικού Διευθυντή. Αυτό θα γίνει με διαγωνισμό στο εξωτερικό και νομίζω ότι ο νέος Επίτροπος είπε ότι είναι διατεθειμένος να συζητήσει το θέμα της ανακοίνωσης, της κοινοποίησης, της ε, χειρεύουσας θέσης ε, με τα άλλα θεσμικά όργανα για να είναι βέβαιοι ότι όλοι θα συμφωνούν με την, ε, τον προσδιορισμό των προσόντων του νέου Γενικού Διευθυντή. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι η υπηρεσία συνεχίζει να λειτουργεί σύμφωνα με τους ε, ε, κανόνες που υπάρχουν και ότι θα επιταχύνουμε την αναζήτηση νέου Γενικού Διευθυντή. Και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δε θα συμμετέχουν στην απόφαση για τα κριτήρια και το προφίλ του νέου Γενικού Διευθυντή και ο διορισμός του νέου Γενικού Διευθυντή θα γίνει σύμφωνα με διοργανική διαδικασία. Τρίτον, για την σύσταση της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων. Πολλή συζήτηση έχει γίνει, ίσως όχι με αυτή την Επιτροπή, αλλά με το Κοινοβούλιο, ναι. Έγιναν πολλές συζητήσεις με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και μέλη του Κοινοβουλίου που εργάστηκαν πάνω στη συνθήκη και στην Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων ειδικότερα. Είναι περίπλοκο το θέμα γιατί θα πρέπει διάφορο, διάφοροι ε, ε, υπάλληλοι να συνεργαστούν και να δημιουργηθεί κάτι καινούργιο και μοναδικό, αλλά νομίζω ότι ακολουθήσαμε τη σωστή προσέγγιση, διότι είπαμε ότι πρώτα πρέπει να επεξεργαστούμε και να καταλήξουμε στο τι θέλουμε να κάνει αυτή η υπηρεσία εξωτερικών δράσεων και μετά θα δούμε αν χρειαστεί ενδεχομένω αλλαγή των κανόνων για να μπορεί να παίζει το ρόλο τη όπω πρέπει η υπηρεσία αυτή. Τώρα αυτό που κάνουμε και αυτό θα υποβληθεί βέβαια θα έρθει και στο Κοινοβούλιο είναι διάφορα πράγματα. Θα, ο ύπατος, η εκπρόσωπος θα υποβάλει πρόταση μετά από διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο και με την έγκριση της Κομισιόν για να συσταθεί, να δημιουργηθεί υπηρεσία. Πιστεύουμε ότι θα καταστεί αναγκαίο να τροποποιηθεί ο δημοσιονομικός κανονισμός ώστε η Κομισιόν να υποβάλει επίσημη πρόταση η οποία θα υποβληθεί σε το χρόνο στο Κοινοβούλιο και πιστεύουμε επίσης ότι θα πρέπει να αλλάξουμε το κανονισμού τους κανονισμούς για το προσωπικό. Παράδειγμα, οι υπάλληλοι της Κομισιόν δεν μπορεί να παίρνουν οδηγίες από κάποιον που δεν είναι στην Κομισιόν. Εντάξει, ως εδώ λειτουργήσε το σύστημα, όμως στο μέλλον θα πρέπει για εκείνους που εργάζονται για την Κομισιόν να δέχονται και από την ε, Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων. Άρα πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός του προσωπικού για να μπορεί να γίνεται αυτό. Γιατί η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων δεν θα είναι επισήμως μέρος της Κομισιόν. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για το ότι πρέπει να τροποποιηθεί. Τώρα ακόμα προσπαθούμε να επεξεργαστούμε ακριβώς ε, ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες της ε, υπηρεσίας εξωτερικών δράσεων. Νομίζω ότι είναι σαφές και λογικό φαίνεται δηλαδή είναι για τις δικές της διοικητικές δαπάνες και στο Ινακρόαση με το Κοινοβούλιο είπα ότι εκπρόσωπος ήδη κατέστησε σαφές ότι δέχεται απόλυτα ότι θα είναι υπόλογη στο Κοινοβούλιο για τις διοικητικές αυτές δαπάνες και το χειρισμό τους. Πιστεύουμε ότι καλό θα ήταν για τις επιχειρησιακές δαπάνες, υπηρεσίες και εσωτερικών υπηρεσιών να παραμείνει στην Κομισιόν η οποία θα ε, υλοποιεί τα προγράμματα για τη βοήθεια στον προϋπολογισμό. Αν γίνει αυτό στο τέλος και θα πρέπει να συζητήσουν όλα τα θεσμικά όργανα, η Κομισιόν θα παραμείνει υπόλογη σε εσά για τη συντριπτική πλειοψηφία των δαπανών, των πραγματικών δαπανών της Ένωσης. Αυτές είναι κάποιες ιδέες που τώρα διαμορφώνονται. Πιστεύω ότι θα είναι δυνατόν μέσα σε εβδομάδες, σε λίγες εβδομάδες μάλιστα, θα είναι δυνατόν η Κομισιόν να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού και μια άλλη για την τροποποίηση των κανονισμών που διέπουν το προσωπικό. Και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα συμμετέχουν στη συζήτηση που είναι απαραίτητη για να συμφωνήσουμε επί της αρχιτεκτονικής υπηρεσίας εξωτερικών ε, δράσεων. Θέλουμε λοιπόν να υποβάλουμε προτάσεις που θα δώσουν δυνατότητα να γίνουν διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις για αυτή την αρχιτεκτονική και το, την υπηρεσία. Ευχαριστώ. Έχουμε 20 λεπτά για 5 ερωτήσεις και 5 απαντήσεις στις 5 ε, και 40 θα έχουμε ολοκληρώσει το θέμα αυτό. Η κυρία Γιάλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την ε, Γενική Γραμματεία για όλες αυτές τις συμπληρωματικές πληροφορίες που μας δίνει. Συγκεκριμένα, θέλω να ρωτήσω την ε, Γενική Γραμματέα το εξή. όσον αφορά την τροπολογία που προβλέπετε του δημοσιονομικού κανονισμού λόγω της νέας αυτής δομής της υπηρεσία για την εξωτερική δράση. Σας ρωτώ το εξή πιστεύετε ότι θα πρέπει να αλλάξουμε κάτι το οποίο μέχρι στιγμής έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Δηλαδή, ε, η Επιτροπή ολοκληρώνει και υλοποιεί προγράμματα και δεσμεύσει που ξεπερνούν τις δημοσιονομικές προοπτικές, π.χ. Γαλιλαίο, και από την άλλη Όσον αφορά τα πολιετή προγράμματα, αυτά αποτελούν αντικείμενο ελέγχου από το συνέδριο σε αιτήσια βάση. Να λοιπόν, ε, με, ε, ε, ε, αυτές είναι οι εξηγήσεις που μας δίνουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής όσον αφορά συγκεκριμένα επίπεδα σφαλμάτων συγκεκριμένες χρονιές. Ρωτώ, δεν προβλέπετε μηχανισμούς διόρθωσης αυτής της κατάστασης. Επίσης, όσον αφορά την εξωτερική δράση. Ήδη μας είπατε τι θα σκοπεύετε να κάνετε. Αλλά θα ήθελα να μάθω το εξής. Σε αυτή την αλλαγή του δημοσιονομικού κανονισμού θα μπορούσαμε εκτός από τα άρθρα, με βάση τα άρθρα 110 έως 118, ένα συγκεκριμένο μηχανισμό ελέγχου κρίσης. Γιατί εδώ προβλέπονται ορισμένε εξαιρέσει σε περίπτωση κρίση, αλλά δεν βλέπουμε μια συγκεκριμένη διαδικασία, ένα συγκεκριμένο μηχανισμό καλά καθορισμένο, ε, γύρω από τον οποίο να υπάρχει συνένεση. Και τέλο, όσον αφορά την Όλαφ, η Επιτροπή Επαγρύπνηση και Εποπτεία σίγουρα μα εξέφρασε τι ανησυχίε τη και εμεί ανησυχούμε, κυρία Γενική Γραμματέα. Δηλαδή, η Όλαφ είναι ένας πολύ, ε, ε, ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Λέω λοιπόν Πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση, πώ θα αντικατασταθεί ο κύριο Μπρένερ, αλλά δεν νομίζω ότι ε, αυτό έχει να κάνει μόνο με την άποψη ενό θεσμού. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ξέρει τι θα γίνει του επόμενου μήνε και τι αποφάσει θα ληφθούν ε, σε αντικατάσταση του κυρίου Μπρένερ. Γιατί ο εσωτερικό μηχανισμό αντικατάσταση τη Όλαφ δεν χαρακτηρίζεται από μια σαφή ιεράρχηση, είναι κάτι τελείω εσωτερικό. Μα εμεί θέλουμε περισσότερε πληροφορίε ζήτημα αυτό. Θέλουμε να μάθουμε τι ακριβώ γίνεται. Σα παρακαλώ να απαντήσετε. Thank Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, για την πρώτη σας ερώτηση. Η πρόθεση της Επιτροπής είναι να περιοριστεί η πρόταση ε, για αλλαγή του δημοσιονομικού κανονισμού μόνο σε ό,τι είναι απαραίτητο για τη δημιουργία της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Δηλαδή η επιθυμία όλων είναι να δράσουμε γρήγορα. Κοιτάξτε, πρόκειται ε, για το πιο, αν θέλετε, ορατό σημείο της συνδίκης Λισαβόνας. Άρα λοιπόν Θέλουμε να περιοριστούμε μόνο σε αυτό που σας είπα. Το Μάιο, όπως σας είπα, θα έχουμε προτάσεις για μία, ε, ε μάλλον θα κάνουμε ε, ένα, γενικές προτάσεις για αλλαγή του δημοσιονομικού κανονισμού και θα μεταφέρω και αυτά τα οποία είπατε για τον Γαλιλαίο. Πάντως δεν εντάσσεται στις αλλαγές που αφορούν την εξωτερική δράση. Για το θέμα του ελέγχου των κρίσεων. Δεν ε, έχω απόλυτα ξεκάθαρο στο μυαλό μου Πού, που, ε, ε, ποια ήταν η πρόθεσή σα με την ερώτησή σα, Ναι, σίγουρα, η ε, πρόθεσή μα είναι να έχουμε ταχύ απόκριση σε, σε επίπεδο κρίση. Και ε, εάν εξακολουθήσουμε να έχουμε τι ίδιε αρμοδιότητε, θα έχουμε και τι ίδιε ρυθμίσει ε, λογοδοσία στο Κοινοβούλιο όπω είχαμε μέχρι τώρα. Αν υπάρξει αλλαγή, και, αλλαγή συγγνώμη, και αν η εξωτερική δράση, η υπηρεσία εξωτερική δράση θα είναι υπεύθυνη για μέρο τη δράση ε, που μέχρι στιγμή είχαμε αρμοδιότητα, τότε τα πράγματα θα ρυθμιστούν ε, με άλλο τρόπο. Αυτό μου είναι λιγότερο πιθανό. Όσον αφορά την Όλαφ, επιτρέψτε μου να, σας, να προσπαθήσω να εξηγήσω τι ακριβώ γίνεται σε αυτέ τι ατυχεί περιστάσει όπου ε, έχουμε το θάνατο κάποιου υπευθύνου ή καινή θέση κτλ. Οι κανόνε προβλέπουν ο προσβήτερο στην υπηρεσία να αναλάβει τι ευθύνε μέχρι να υπάρξει ο νέο διορισμό. Και ακριβώ αυτό έγινε στην Όλαφ. Τώρα, ο προσβήτερο είχε ήδη διοριστεί στο παρελθόν από τον κύριο Μπρίνερ ω αντικαταστάτης του. Άρα δεν υπάρχει κενό. Πρέπει να υπάρξει συνέχεια, είναι απαραίτητο και όπω και στι υπόλοιπε υπηρεσίε τη Επιτροπή, όπου απουσιάζει ο γενικό διευθυντή, για οποιοδήποτε λόγο, όχι μόνο λόγω θανάτου, αλλά για άλλου λόγου. Ο πρεσβύτερο ε, αναλαμβάνει, ο, πρε, ο μάλλον. Και σε αυτή την περίπτωση επαληθεύσαμε τι νομικέ υπηρεσίε ότι αυτό ήταν το σωστό ε, και επιβεβαιώσαμε και αυτή την περίπτωση. Τώρα, φυσικά, αυτή δεν είναι μια επιθυμητή κατάσταση ε, μακροπρόθεσμα. Κάθε υπηρεσία χρειάζεται σαφή ηγεσία, ξεκάθαρα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς αποφασίσαμε να επιταχύνουμε τη δημοσίευση της ε, καινής θέσης αυτής. Θα απαιτηθούν όμως κάποιοι μήνες. Πρέπει να γίνει δημοσίευση, ε, να προκήρυξη, να εξετάσουμε του υποψήφιου, να διοργανώσουμε τι συνεντεύξει. Ε, ε, θα πρέπει να έρθω στο Συμβούλιο, στο Κοινοβούλιο. Άρα ε, απαιτείται κάποιο χρόνο. Στο μεταξύ, καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να αφήσουμε την υπηρεσία ακέφαλη. Ακριβώ γι' αυτό ακολουθήσαμε του κανόνε που ακολουθούμε σε όλε τι περιπτώσει, σε όλε τι παρόμοιε περιπτώσει. Η συνέχεια τη υπηρεσία εξασφαλίζεται και θα ξεκινήσουμε την προκήρυξη ε, ώστε να τον πιο γρήγορα. Αλλά όπως σας είπα, η επόμενη Επιτροπή ήδη είπε ότι θα συζητήσει ε, της τη της κενής με τους υπόλοιπους θεσμούς, έτσι ώστε όλοι να είμαστε σίγουροι ότι περιγράφονται σωστά ε, τα προσόντα του υποψηφίου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, κύριε Αντρεάσεν. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, να απαντήσατε στην ερώτηση του κυρίου Λιμπεράσια αλλά ε, θα ήθελα να σας πω ότι δεν ικανοποιήθηκα διότι η Επιτροπή είχε ζητήσει να εξεταστεί ε, ε, να γίνει μια μελέτη σχετικά με τον κώδικα συμπεριφοράς των Επιτρόπων και θα ήθελα ίσως να σας πω ότι είδαν ότι υπήρχαν συγκρούσεις συμφερόντων και ε, έχετε διατυπιστώσει τέτοιες συγκρούσεις συμφερόντων. Η δεύτερη ερώτησή μου αναφέρεται εις τους κανόνες που διέπουν τις προσλήψεις προσωπικού. Είπατε ότι θα ενημερώσετε τον ε, εσωτερικό κανονισμό όσον αφορά το προσωπικό διότι έχουμε ήδη ε, το 2006 καταρτήσει μία μελέτη ε, για τις ε, ε, αναφορές και είχαμε ζητήσει από την Επιτροπή να μας, να μας ενημερώσει για τα θέματα αυτά των διαρροών. Ναι, γνωρίζω το θέμα, γνωρίζω τις συστάσεις σας και όποτε η Επιτροπή αναθεωρήσει τον κώδικα συμπεριφοράς θα το συμβουλευτούμε. Γνωρίζω επίσης ότι πρέπει να ζητούμε από αυτούς οι οποίοι αισθάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά με το σύστημα να το λέγουν. Χωρίς όμως να αισθάνομαι ότι χρειάζεται να αλλάξει ο εσωτερικός κανονισμός για το προσωπικό για να το επιτύχουμε. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας κώδικας ηθικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και να υπάρχουν σε όλες ε, τις ε, ε, διευθύνσεις συνεδριάσεις όπου να τονίζεται ότι όποιος αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά πρέπει να το επισημαίνει. Ξέρω ότι συνήθως προσπαθεί κανείς να βελτιώσει το κλίμα κατά τρόπον ώστε κάποιος να μπορεί να επιβραβεύεται σε περίπτωση που επαγρυπνεί και αυτό είναι πιο αποτελεσματικό από το να αλλάξουμε ε, τους κανόνες και ο εσωτερικός κανονισμός για το προσωπικό δεν ε, χρειάζεται γενική αναμόρφωση μόνο σε συγκεκριμένα σημεία. Δεν νομίζω δηλαδή ότι όλα πρέπει να αναθεωρηθούν. Θα δείτε ότι υπάρχει θετική ενθάρρυνση για το προσωπικό και ξεκινάει και από τον πρόεδρο. Εάν κάποιος ε, διαπιστώσει ή υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά πρέπει αμέσως να ενημερώσει την διοίκηση. Ευχαριστώ. Έχουμε 10 λεπτά για τρία ερωτήματα. Παρακαλώ λοιπόν να είστε πολύ σύντομος. Ο κύριος Κάλφη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επανέλθω στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί πολύ στο μέλλον. Είπατε ότι υπάρχει ένα τμήμα το οποίο έχει ε, ε, συγκεκριμένες αρμοδιότητες όπου η ύπατος εκπρόσωπος θα ε, είναι υπεύθυνη για τα διοικητικά έξοδα και ε, ο Επίτροπος για τα λειτουργικά. Αλλά έχει ε, σταθεί σχεδόν αδύνατο να μπορέσει κανείς να κάνει ένα καλό διαχωρισμό μεταξύ διοικητικών, διαχειριστικών και επιχειρησιακών δαπανών. Οπότε πολύ φοβάμαι ότι θα δημιουργηθούν ακόμη περισσότερα προβλήματα. Ποιο είναι το σύστημα οικονομικού ελέγχου το οποίο θα καταρτήσετε. Θα αλλάξετε όλο το σύστημα στην νέα υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Θα είναι ανεξάρτητο από την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Και πώς θα εξασφαλίσετε τη συνεκτικότητα και τον έλεγχο αυτού του οικονομικού συστήματος. Και μια άλλη παρατήρηση σχετική με αυτή εφόσον ορισμένοι επικεφαλής των αντιπροσωπιών πλέον του να είναι οι υπόλογοι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι υπόλογοι και προς τα ταμεία που τους χρηματοδοτούν πώς πιστεύετε ότι θα μπορέσουν να συνδυάσουν την ε, υποχρέωση που θα έχουν έναν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αυτή που θα έχουν έναν των ταμείων και τέλος θα ήθελα ε, να ρωτήσω κάτι ακόμη. Ε, ε, μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η αναπτυξιακή πολιτική την οποία έχει αναλάβει η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές. Ε, θα ξεκινήσω αυτά που έχω να πω λέγοντας ότι τίποτα δεν είναι τελεσίδικο. Απλώς είναι ιδέες τις οποίες εξετάζουμε και κοιτάζουμε να δούμε ποιο μείγμα ιδεών θα επιλεγεί από την το εκπρόσωπο για ε, τα θέματα που θα διεκπεραιώνει. Θα θέλαμε να ψάξουμε να βρούμε έναν τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να εκτελεί πολλά καθήκοντα για την υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης το οποίο θα ήταν οικονομικό για τον προϋπολογισμό ε, θα επιτρέψει στην μονάδα εξωτερικής δράσης να μην επεκταθεί θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε το σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα είμαστε αρκετά πιστικοί για να μπορέσουμε ε, να επιτύχουμε την συνεργασία με, το, ε, ε, με την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων και σε οικονομικό τομέα. Δηλαδή να δούμε εάν μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα ABAC που πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνει αν ο ε, επικεφαλής του λογιστηρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να αναλάβει και την υπηρεσία εξωτερικής δράσης αν θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ο εσωτερικός οικονομικός ελεγκτής ή θα χρειαστούν εξωτερικοί ελεγκτές για αυτές τις υπηρεσίες. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες που μας απασχολούν αυτή τη στιγμή όπου δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί κάτι νέο θα μπορέσουμε να οριοθετήσουμε σωστά τις υπηρεσίες και να τις μοιραστούμε. Οι αντιπροσωπείες βέβαια θα είναι στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης αλλά θα μπορεί να υπάρχει και ανάθεση για την δημοσιονομική διαχείριση άρα να είναι υπόλογη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με αυτόν τον τρόπο να εκμεταλλευτούμε μία από τις δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν. Επιπλέον θα υπάρχει συνέχεια και συνέπεια χωρίς να χρειαστεί να αναπτυχθεί ένα νέο σύστημα. Αν όμως δεν υιοθετηθεί αυτό το πρότυπο θα χρειαστεί να σκεφτούμε κάτι άλλο αν και θεωρούμε ότι αυτό θα είναι το πιο οικονομικό και θα επιτρέψει την καλύτερη συνέχεια της, ε, των υπηρεσιών. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να επηρεάζει την ε, διαμόρφωση πολιτική στο μέλλον και η υπεύθυνη για την αναπτυξιακή πολιτική θα είναι αρμόδια για το μέλλον και θα πρέπει να δούμε πού θα γίνεται ο προγραμματισμός των εργαλείων για την ανάπτυξη και αυτό το θέμα δεν έχει ακόμη επιληθεί. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση την κάνω εγώ. Ε, ε, Γενική Γραμματέα και μετά θα τελειώσουμε. Επειδή υπάρχουν, είναι ακόμα πολλές οι απάτες, όπως φαίνεται ιδιαίτερα από τις εργασίες όχι μόνο του, της Όλαφ, αλλά και από το γεγονός ότι το Κεντρολικό Συνέδριο έχει βρει ε, σοβαρές παρατυπίες. Τώρα, ε, όσον αφορά την ενίσχυση του ρόλου της Όλαφ, όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά, θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Ε, ε, τι, ε, ε, πώς βλέπετε το θέμα της προκήρυξης των διαγωνισμών, γιατί υπάρχουν σοβαρές παραβάσεις, όπως ακούσαμε και σήμερα το απόγευμα το ελεκτικό συνέδριο. Και τέλος, πώς βλέπετε το θέμα των κυβερνήσεων και των κρατών μελών όπου καταγράφονται οι περισσότερες περιπτώσεις παρατυπίας και διαφθοράς έναντι των κοινωτικών κονδυλίων, των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Τι σκέφτεστε να κάνετε απέναντι όσον αφορά όλα αυτά τα ζητήματα. Well, Λοιπόν, προφανώς η Όλαφ είναι μέρο τη Επιτροπή, αλλά είναι και ανεξάρτητο οργανισμό. Άρα η ίδια η Όλαφ θα αποφασίσει τι μελέτε απαιτούνται, αν θεωρεί ότι απαιτούνται μελέτε ε, που θα ε, βελτιώσουν τις εργασίες της. Ε, εγώ να σας πω το εξής. Εμείς ως Επιτροπή, όταν βλέπουμε ότι όταν έχουμε να κάνουμε απάντηση που ανακαλύπτει η Όλαφ, να σα πω τι κάνουμε, πώς αντιδράμε. Λοιπόν, σε τακτικά χρονικά διαστήματα ε, έχουμε κάνει όλο και πιο αυστήρου του κανόνες όσον αφορά την προκήρυξη διαγωνισμών και τις ε, συναφείς διαδικασίες όταν ανακαλύπτουμε κάποιε απάτες. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο ε, κάνουμε μετά από την ε, Όλαφ, δηλαδή αφού έχει κάνει τις έρευνές η Όλαφ και έχει ενδεχομένως εντοπίσει επιμέρους υποθέσεις ή αδυναμίες στο σύστημα ελέγχου, τότε εμείς ε, ως Επιτροπή αναλαμβάνουμε δράση για να κάνουμε πιο αυστηρούς κανόνες σε ολόκληρη την ε, Επιτροπή. Εμείς με αυτόν τον τρόπο αντιδρούμε και προσπαθούμε να αντλήσουμε διδάγματα σε περιπτώσεις απατών στο παρελθόν. Δεν συμφωνώ ότι απάτε και παρατυπίε είναι το ίδιο πράγμα. Πρέπει να κάνουμε διάκριση. Όταν έχουμε απάτε, ακόμα και όταν δεν έχουμε απάτε. Αλλά όταν οι έρευνε δείχνουν ότι υπάρχουν αδυναμίε στο σύστημα, τότε προσπαθούμε να απαντήσουμε με συστηματικό τρόπο. Δηλαδή να αλλάξουμε του κανόνε, να του προσαρμόσουμε, να του κάνουμε πιο αυστηρού και αυτό συνολικά στην Επιτροπή και να ε, διδαχθούμε από την εμπειρία μα. Τώρα, όσον αφορά ε, την αντιμετώπιση των κρατών μελών Διακόπτη μιλήτρια. Και εδώ νομίζω ότι τα πρόσφατα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, έχουμε εντείνει το διάλογο σε θέματα ελέγχου και, ε, ε, και διοργανώνουμε σε τακτικά χρονικά διαστήματα εργαστήρια, για παράδειγμα, τα κράτη-μέλη, για να του βοηθήσουμε να βελτιώσουν το σύστημά του. Νομίζω ότι στην τελευταία ανάλυση ε, το, το, το, το όλο έγκυται σε μια συμπεριφορά ραβδιού και καρότου. Δηλαδή, από τη μια κάνουμε πιο αυστηρού του ελέγχου, και από την άλλη ε, από τη μια προσπαθούμε να τους πείσουμε και από την άλλη έχουμε αυξήσει την προσφυγή μα ε, στα ε, συστήματα ανάκτησης που βεβαίω αποτελούν έναν τρόπο προστασίας των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωση και από την άλλη με τον τρόπο αυτό κάνουμε και τα κράτη-μέλη να καταλάβουν ότι απαιτείται να λάβουν μέτρα ενίσχυση των δικών του ελέγχων. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστούμε κύριε Αντέη. Έχουμε τώρα τον Αντιπρόεδρο κύριο Πιτέλα και τον Γενικό Γραμματέα Κλάους Βέλλα και με αυτόν τον τρόπο πάμε στο θέμα 9, απαλλαγή 2008, Γενικός Προϋπολογισμός ε, Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συγκεκριμένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στον κύριο Ιωάννη Σαρμά, εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, Προηγουμένως παρενέβην και είπα ότι το ελεγκτικό συνέδριο για το κεφάλαιο 11 έχει εκδώσει ένα συλλογικό συμπέρασμα για όλα τα θεσμικά όργανα χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένα στο Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε κάποιο άλλο θεσμικό όργανο. Στο κεφάλαιο 11 καλύπτονται όλα τα θεσμικά όργανα. Παρ' όλα αυτά θα δείτε σε τέσσερις κατηγορίες ε, ε, πληροφοριών τα ε, συμπεράσματά μας όσον αφορά το Κοινοβούλιο. Και εδώ αναφερόμαστε καταρχήν εις τις συναλλαγές σε επίπεδο του Κοινοβουλίου που δεν μας έχουν δημιουργήσει οποιαδήποτε ανησυχία. Δεν υπάρχουν δηλαδή ουσιαστικά λάθη στις συναλλαγές του Κοινοβουλίου και όσον αφορά το σύστημα εσωτερικού ελέγχου έχουμε μία θετική αξιολόγηση. Τώρα, όσον αφορά τις συγκεκριμένες, τους συγκεκριμένους ελέγχους ε, είχαμε βρει μία πληρωμή η οποία έγινε ως προκαταβολή και ήταν παράτυπη αλλά η απάντηση του Κοινοβουλίου μας ικανοποίησε πλήρως. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σχετικά με το θέμα αυτό. Ε, όσον αφορά τις εσωτερικές μας τώρα παρατηρήσεις έχουμε τέσσερις τομείς. Πρώτον, τα θέματα, το θέμα του πολλαπλασιαστή που εφαρμόζεται στο Κοινοβούλιο διότι το Κοινοβούλιο δεν, δεν εφαρμόζει με τον ίδιο τρόπο το συντελιστή πολλαπλασιασμού και υπάρχει μία υπόθεση η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και όταν αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα έχουμε κάποια λύση. Μέχρι τότε το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να εφαρμόζει ε, και να ερμηνεύει τον ε, κανονισμό με τον ίδιο τρόπο που κάνει και τώρα. Ε, το δεύτερο αναφέρεται εις την καταποκοπή καταβολή των εξόδων της διανυκτερεύσεως για τα τρία σημεία εργασίας του Κοινοβουλίου. Δεν υπάρχει δηλαδή με μονομένη η ανάλυση των εξόδων αποστολή όπως εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε να υποχρεωθεί το Κοινοβούλιο αντιθέτως για λόγους οικονομιών και για άλλους λόγους που μας εξηγεί το Κοινοβούλιο στην απάντησή του υπάρχει ένα ποσό κατά στο σημείο αυτό μπορούμε να πούμε ότι κάναμε μία προσπάθεια για να συνεννοηθούμε. Αλλά το θέμα δεν έχει λυθεί. Το, Ευρω... το ελεγκτικό συνέδριο περιμένει ή να αλλάξει ο εσωτερικός κανονισμός ή το δημοσιονομικός κανονισμός, δηλαδή σε υψηλό επίπεδο μία ρύθμιση που να επιτρέψει να λυθεί το θέμα. Όσον αφορά το τρίτο θέμα που είναι οι αποζημιώσεις προς τους ευρωβουλευτές βουλευτές έχουμε κάνει σημαντικές προοδούς διότι εδώ αναφερόμασταν εις, ε, τις, ε, στα διάφορα επιδόματα του προσωπικού από το 2004 2007 και βλέπουμε ότι το Κοινοβούλιο προχωρά στον έλεγχο των διαφόρων ε, δικαιολογητικών που προσκομίζουν οι ευρωβουλευτές. Και τέλος όσον αφορά τα ε, στις επιπρόσθετες δαπάνες υπάρχει μεγάλη βελτίωση διότι το συνέδριο δημοσιεύει ε, το αποτέλεσμα συγκρίνουμε με το αποτέλεσμα του συνταξιοδοτικού ταμείου έχουν ε, ληφθεί μέτρα για να μειωθεί το έλλειμμα και καλέσαμε το κοινοβούλιο να κάνει μία αντασφαλιστική μελέτη για να δει ποσο ποιες θα είναι μακροπρόθεσμα οι επιπτώσεις αυτού του θέματος. Ωραία. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον Αντιπρόεδρο κύριο Πουτέλα, ο οποίο είναι υπεύθυνο όσον αφορά τον, ε, το θέμα αυτό του ισολογισμού των ε, ε κοινοτικών οργάνων. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εξ ονόματο του συναδέλφου Βιντάλ Κουάντρα, με τον οποίο συνεργαζόμαστε στη διαχείριση ε, του, του θέματο αυτού του, που, και των ευθυνών των αμβλητών του προπολογισμού. Επιτρέψτε μου να σα χαιρετήσω όλου, τον εισηγητή για την απαλλαγή, του αντιπρόεδρου τη Επιτροπή, Ελέγχου Προπολογισμού, όλους τους συναδέλφους, ε, μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού, με πολλούς από τους οποίους είχα την ε, ευχαρίστηση να, με πολλούς από τους οποίους είχα την ευχαρίστηση να συνεργαστώ και στο παρελθόν. Πρέπει να σας πω ότι είχα την τιμή να είμαι μέλος της Επιτροπής σας. Στην αρχή της ε, θητείας μου στο Κοινοβούλιο πριν από 10 χρόνια περίπου και διδυρώ μια ιδιαίτερα θετική ανάμνηση από αυτή τη θητεία. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί σήμερα ε, συνοδεύομαι από τον Γενικό Γραμματέα, τον Κλάους Βέλ, από τον κύριο Ρόμπερτ Γκάλβιλ και από τον κύριο Ιωάννη Σαρμά ο οποίος ε, ε, είναι μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου και ο οποίος μόλις ε, μας ανέπτυξε τις δικές του απόψεις, την αξιολόγησή του και την κρίση του. Και χαίρομαι ιδιαίτερα και αισθάνομαι ιδιαίτερη επιφαρηφάνεια, γιατί όσον αφορά τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, δεν αναφέρθηκαν θετικά σχόλια Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να ζητάμε από τους άλλους να είναι διαφανείς ε, και ε, να έχουν ορθή διαχείριση των δαπανών τους αν δεν είμαστε εμείς που θα δώσουμε το παράδειγμα. Και νομίζω ότι πραγματικά μέσα από την πάροδο όλων αυτών των χρόνων δείχνουμε ότι όλο και περισσότερο μας χαρακτηρίζει η διαφάνεια και ότι έχουμε φτάσει σε κάποια πρότυπα ε, όσον αφορά τις δαπάνες και την ορθότητα των δαπανών τα οποία είναι σημαντικά. Όπως τα ξέρετε πολλοί από εσάς είναι ο δεύτερος χρόνος που ένας αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου συμμετέχει στην ακρόαση για την απαλλαγή του προπολογισμού και νομίζω ότι αυτό ε, θα πρέπει να το δείτε στην οπτική γωνία της καλής σχέσης και τη στενή συνεργασία του Προεδρείου με την Επιτροπή Προϋπολογισμού και με την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Ο στόχο τη σημερινή συζήτηση είναι να αναλύσουμε την κατάσταση του προπολογισμού για το 2008, για το οικονομικό έτο 2008 και να ε, ε, δούμε τι αποφάσει ε, του Προεδρείου που προφανώ είχαν επιπτώσει στον προπολογισμό. Τόσο διότι οι πιστώσει ήδη εντάσσονται σε, ένα, σε, μία γραμμή, σε ένα κονδύλιο του προπολογισμού και γιατί η προπολογιστική αρχή προέβη σε μεταφορά πιστώσεων για τη, για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων γραμμών του προπολογισμού. Να σα δώσω κάποια γενικά στοιχεία. Συνοψίζοντα, όσον αφορά το επίπεδο των οριστικών πιστώσεων, ήταν 1.425.517 ευρώ. Όσον αφορά το επίπεδο των ανάληψης υποχρεώσεων, 1.401.900 ε, που αποτελεί το 97% των οριστικών πιστώσεων. Το σύνολο των πληρωμών ένα δις 200 που είναι το 97% των ε, πιστώσεων που είχαν αναλυφθεί, το επίπεδο των αυτόματων μεταφορών που είχαν καταληφθεί το 2008 και πληρώθηκαν το 2009, 196, 133, 738, ενώ οι μη αυτόματες ε, μεταφορές το 2009 8.315-729 ε, ευρώ. και ε, πρέπει να πούμε ότι ε, αυτά τα αριθμητικά στοιχεία δείχνουν ότι χαρακτηριζόμαστε από ιδιαίτερη διαφάνεια και δείχνουν ότι ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός ο τρόπος αντιμετώπισης των δαπανών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να πούμε ότι η εκτέλεση ε, ήταν της τάξης του 97%. Τώρα, να πάμε στην παράθεση. Ξέρω ότι όλα αυτά είναι κάπως κουραστικά και βαρετά και σας ζητώ συγγνώμη, αλλά είμαι αναγκασμένος να το πράξω γιατί θα πρέπει να προβώ σε απολογισμό όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν από το Προεδρείο του Κοινοβουλίου ε, και γιατί από τις αποφάσεις αυτές ε, απορρέουν οι δαπάνες. 14 Πρώτου 2008. Το Προεδρείο, όπως κάθε χρόνο, αποφασίζει προσωρινό ποσό για την υποστήριξη ε, του, του οργανισμού των πρώην ε, μελών του Κοινοβουλίου. 251.000 ευρώ είναι το ποσό αυτό. Επίσης, το Προεδρείο ε, διαβουλεύει, συζητά χωρί συζήτηση και εγκρίνει την πρόταση ε, της συνδιάσκεψη των Προέδρων όσον αφορά τις πιστώσεις για την 4.000 γραμμή για 2007 ε, προϋπολογισμός λειτουργίας των πολιτικών ομάδων. 57 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Επίσης, το Ιανουάριο του 2008 εγκρίνει την πρόταση των κοσμητόρων για αύξηση των δαπανών των βοηθών των βουλευτών 1.418 ευρώ για κάθε βουλευτή ξεκινώντας από την 1η Πρώτη του 2008. 13 ε, δις ευρώ σημαίνουν όλα αυτά στον προπολογισμό 18 Δευτέρου 2008 εγκρίνεται ε, η, η σύσταση που αφορά ε, τα πολιτικά κόμματα στο επίπεδο Ευρώπης 10.339.000 ευρώ. Επίσης εγκρίνεται η πρόταση αγοράς ε, του κτηρίου ε, ε, στο Λονδίνο για εγκατάσταση του ενημερωτικού γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνολικό κόστος συν εργασίες 35 εκατομμύρια ευρώ. στο προπολογισμό ακριβώς το ποσό που εγγράφεται είναι 35 εκατομμύρια ευρώ. Υπογραμμίζω ότι αυτή η αγορά, όπως και άλλες, μας επέτρεψε να εξοικονομήσουμε από τις δαπάνες σημαντικά, σημαντικό ποσό χρημάτων γιατί ε, αν εξακολουθούσαμε να νοικιάζουμε θα πληρώναμε συν 17 ε, εκατομμύρια μέσα στα 20 χρόνια. Το, ε, το Προεδρείο επιβεβαιώνει την απόφασή του ανα, αναδιάρθρωση των αιθουσών στο Στρασβούργο για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες διερμηνίας σε 20 αίθουσες. 1,2 εκατομμύρια ευρώ, κόστος των εργασιών κτλ. Ε, όσον αφορά την αύξηση των γλωσσών. Λοιπόν, ε, αυτό ε, είναι μια απόφαση που εγκρίθηκε το Μάιο 2008. Το Μάρτιο 2008 το Προεδρείο μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα για την κατάσταση που αφορά το ενίκιο του κτηρίου στις Βρυξέλλες ενέκρινε την υπογραφή σύμβασης. E ε, ε, ναι, έχουν δίκιο οι λέει ο μιλητή. Πραγματικά και οι συνάδελφοι. Μιλάω πολύ γρήγορα και δίνω στοιχεία. Όλα αυτά ε, έχουν συνέπειε στον προπολογισμό και χρηματοδότηση από το υπόλοιπο του υπερπολισμού 2007 18,5 εκατομμύρια ευρώ. Εγκρίθηκε η συγκεκριμένη συναλλαγή 8 Μαρτίου 2008. Το ε, Προεδρείο εγκρίνει για πέντε χρόνια ενοικίαση αίθουσας πληροφορικής για, 200, μια αίθουσα 250 τετραγωνικά. 396.000 ευρώ είναι το ποσό στον προπολογισμό. 9 Τετάρτη 2008 το Προεδρείο εγκρίνει τη χρηματοδότηση για το αρχείο των πρώην βουλευτών. 7 Πέμπτου 2008 ε, το Προεδρείο εγκρίνει την πρόταση των κοσμητόρων και του Γενικού Γραμματέα με στόχο την τροποποίηση ε, της εισόδου επισκεπτών στο Στρασβούργο και εγκατάσταση ανελκυστήρα ε, που να επιτρέπει τη σύνδεση με το πάρκιν. Πως, ε, ποσό στον 900.000 ευρώ ε, συμπεριλαμβανομένων και των μελετών στο ποσό αυτό. Αυτή η απόφαση δεν αφορά τον προπολογισμό 2008, δεδομένου ότι ε, οι μελέτες, οι δημοπρασίες κτλ. εκτιμήθηκε σε 18 μήνες. Οι, οι απαραίτητε επιστώσει θα προβλεφθούν στο σχέδιο προπολογισμού 2009. Αποφασίζει το Προεδρείο να φιλοξενήσει την Παγκόσμια Συνδιάσκεψη του 2008 για το ηλεκτρονικό κοινοβούλιο. Το Νοέμβριο του 2008 διοργανώνεται από κοινού η συνδιάσκεψη με το Παγκόσμιο Κέντρο ε, για την πληροφορική και σε συνεργασία με την ε, Διακοινοβουλευτική Ένωση. 323 η γραμμή του προπολογισμού, όπου αναφέρονται τα απαραίτητα κονδύλια και το ποσό είναι 141.000 ευρώ. Το Προεδρείο επίσης εγκρίνει την απόφαση για ε, που αφορά τα πρώην μέλη του Κοινοβουλίου. Ε, έχουμε το δημοσιονομικό δελτίο και το ποσό, το οριστικό ποσό επιχορήγησης είναι 130.000 ευρώ. 6 Ιουνίου 2008 εγκρίνεται η προσαρμογή του Γραφείου Ενημέρωσης του Κοινοβουλίου και Πληροφορίας ε, σχετικά με το Κοινοβούλιο στο Μιλάνο. 149,53 ευρώ. 149.530 ευρώ η επιπτώση στον προπολογισμό. Λοιπόν, στη συνέχεια εγκρίνεται ομόφωνα ε, η, η διεύρυνση του κτηρίου Αντενάουερ στο Λουξεμβούργο με επίπτωση στον προπολογισμό μηδενική. Γιατί? Γιατί η απόφαση δεν έχει επιπτώσει στο συνολικό κόστος του ε, έργου. Η Επιτροπή Προπολογισμού έδωσε τη γνώμη τη με βάση τον δημοσιονομικό κανονισμό. Το Προεδρείο επίση έλαβε την απόφαση μετά ε, από συγκεκριμένη πρόταση για το κτίριο Big West στο Λουξεμβούργο για τις εργασίες ε, διεύρυνσης και του κτιρίου CAD και την ε, μερική εκένωση του συγκεκριμένου κτιρίου. Πάλι δεν έχουμε επιπτώσει τον προπολογισμό για το 2008. Για το 2009 1.274.705 ε, ε, εγγράφησαν στον προπολογισμό. Επίση, η 7 Ιουλίου 2008 το Προεδρείο ενέκρινε την απόφαση για ε, επιχορήγηση των πολιτικών σχηματισμών σύμφωνα με την πρόταση του Γενικού Γραμματέα 4.268.630 ευρώ οι επιπτώσεις. Το Προεδρείο εγκρίνει την σύναψη ε, σύμβασης μίσθωσης για ε, κτίριο στο Βουκουρέστι για να υπάρξει το, ο οίκος της Ευρώπης ε, στη Ρουμανία. 433.603 ευρώ είναι το ποσό στον προπολογισμό. Το Προεδρείο επίσης εγκρίνει την απόφαση για τα πολιτικά κόμματα και εγκρίνει τελική έκθεση ε, ποσό ε, οριστικής επιχορήγησης, το οποίο ε, θα ε, μοιραστεί. Επίπτωση στον προπολογισμό 1.623.456 ευρώ. Το Προεδρείο στη συνέχεια εγκρίνει την απόφαση για τις πολιτικές ομάδες, ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες, λαμβάνει υπόψη και σημειώνει τα έγγραφα και τους τελικούς ενοποιημένους λογαριασμούς των μη εγγεγραμμένων και των πολιτικών κομμάτων στο εγκρίνει τους στο ΕΛΚ το ποσό που, αφορούν, ε, που αφορά για τα 2005 έως 2007 ε, κόστος προσωπικού το οποίο εγγράφηκε χωρίς να πρέπει μετά την 31η Ιανουαρίου 2008. Εξετάστηκαν διάφορα ποσά και αναφέρεται το αντίστοιχο ποσό επίπτωση στον προπολογισμό. Επίσης, στη συνέχεια, το Προεδρείο επιτρέπει την υπογραφή σύμβασης πώλησης ε, για το, ε, ε, σε σχέση με το γραφείο στη Βιέννη. 27.683.432 ευρώ και υπήρξε ε, ένα αίτημα μεταφοράς το οποίο εγκρίνεται στις 18 2007. Πρόκειται δηλαδή για πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από τον προπολογισμό 2007. 3 Σεπτεμβρίου 2008. Το Προεδρείο αποφάσισε να παρατείνει ε, την ε, ενοικίαση του κτίριου στο Λονδίνο. Queen Anne Gate μέχρι να ε, έχουμε τα νέα κτίρια για το Γραφείο Ενημέρωσης υπό τι εξή προϋποθέσεις. Παράταση για δύο χρόνια μέχρι το Μάρτιο του 2011 ε, με δυνατότητα αποχώρηση μετά από 18 μήνες μετά από προειδοποίηση τριών μηνών. 382.500 ευρώ το χρόνο. 704.390 ε, το ποσό στον προπολογισμό που καταλογίζει 2009. 8 Δεκάτου 2008 ε, το ε, Προεδρείο αποφασίζει την υπογραφή σύμβασης για το κτίριο Βίρτς για 15 χρόνια. Καμία επίπτωση του προπολογισμού του 2008 και με αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομήσουμε 400.000 ευρώ το χρόνο. 17 11 2008 το ε, Προεδρείο για ε, ε, συμπληρωματικούς οικονομικούς πόρους και για τη χρηματοδότηση της ενημερωτικής εκστρατείας για το 2009 αποφασίζει τέσσερα, την πίστοση 4 εκατομμυρίων ευρώ στο 2008 και υποδι υποδεικνύεται να υπογραφεί η μεταφορά μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού σύμφωνα με τη διαδικασία που γνωρίζουμε. 4 εκατομμύρια ευρώ επίπτωση στον προπολογισμό. Η Επιτροπή Προπολογισμού έδωσε τη γνώμη τη επειδή ε, πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα, όπως ε, ανέφερε και ο Πρόεδρος και η Επιτροπή ε, Προπολογισμού, ενέκρινε το ποσό αυτό. 19 του 2008 εξετάζεται από το Προεδρείο την πρόταση υπολείπων από τον προηγούμενο προπολογισμό. σημειώνει το στάδιο εκτέλεσης του προπολογισμού. σημειώνει και λαμβάνει γνώση την πρόταση του Γενικού Γραμματέα, την κατάσταση αυτή και αποφασίζει την επανακατανομή με τη μορφή μεταφοράς 2 εκατομμυρίων ευρώ στον προπολογισμό 2008 ε, τη Ευγενική Διεύθυνση ΚΟΜ έτσι ώστε να υπάρξουν περαιτέρω πιστώσει για την διαδικασία ενημέρωση και εξτρατεία ενημέρωση για την ενόψη τη προεκλογική εκστρατεία 2009. 6 εκατομμύρια ευρώ ε, στη γραμμή 4.000 για τις ενημερωτικές δράσεις των πολιτικών ομάδων. Τα υπόλοιπα ε, θα είναι διαθέσιμα τα, τα υπόλοιπα τα διαθέσιμα από την 1η 1η 2008 θα επιστραφούν στα κράτη-μέλη. 8 εκατομμύρια επίπτωση στον προπολογισμό. 3 το 10 του 2008 το Προεδρείο εγκρίνει αύξηση της αποζημίωσης των δαπανών των Ευρωβουλευτών για 2009 3,7%. Καμία επίπτωση στον προπολογισμό του 2008. 15 του 2008 έγκριση της ε, χρηματοδοτικής συνεισφοράς ε, στην ε, ε, Ένωση Μελών του Κοινοβουλίου 140.000 ευρώ. Στη συνέχεια ορίστηκε το ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς στην, στην οργάνωση των πρώην βουλευτών 170.000 ευρώ, καμία επίπτωση στον προπολογισμό για το 2008, γιατί το μέτρο είναι λειτουργικό από το 2009. Το Προεδρείο επίση αποφασίζει ότι το όριο του 50% που προβλέπεται στα άρθρα 216 και 292 του κανονισμού που αφορά τη χρησιμοποίηση των πιστώσεων τη ε, γραμμή του περιβολισμού 4.000 δεν αφορά τι συμπληρωματικές πιστώσει των 6 εκατομμυρίων ευρώ που, αποφάσισε, που αποφάσισε να δώσει στη συνεδρίασή του στις 19 Νοεμβρίου του 2008. Και κατά συνέπεια τα ποσά αυτά τα συμπληρωματικά μπορούν να μεταφερθούν ε, στο ακέραιο στο 2009. Αποφασίζει επίση ότι οι ομάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πιστώσεις αυτές πνευματικές μέχρι το τέλος του Μαρτίου του 2009. Το 2008 το Προεδρείο αποφάσισε εξάλλου ε, ε, ε, σε μία σειρά από εγκρίσεις, περίπου 130, για συνεδριάσεις κτλ. Και άλλα μικροποσά. Μιλάμε για, χιλιάδες, για μερικές χιλιάδες ευρώ, έτσι, δεκάδες χιλιάδες που να μην σας τα παραθέσω όλα αυτά, διαβάστε τα αν θέλετε. Ε, ε, ε, και για μένα έτσι, γιατί, όχι τόσο για εσάς, γιατί ε, ε, και εγώ κουράστηκα και τώρα, εντάξει αυτά είναι σήματα. Μην χάνουμε το χρόνο μας, έχουμε σοβαρά ζητήματα. Σας ζητώ συγγνώμη, ε, ευχαριστώ που με ακούσατε, σας ζητώ συγγνώμη για αυτή την ε, μονότονη και βιαστική παράθεση αριθμητικών στοιχείων, αλλά όφιλα να το κάνω, ε, από τη θέση μου ε, όφιλα να το πράξω και θα απαντήσω Γενικό Γραμματέα σε όλα σας τα ερωτήματα. Εμείς σας ευχαριστούμε. Πριν δώσουμε το λόγο στο Γενικό Γραμματέα, να δώσω ε, το λόγο στον κύριο Ρόμπερτ Γκάλβιν που εξετάζει τους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχετε το λόγο. Ε, κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής, καταρχήν ε, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ε, δυνατότητα που μου δίνετε να παρουσιάσω την ετήσια έκθεση του 2008. Στις 30 Ιουλίου κατέληξα μετά από διαβουλεύσεις με τον Γενικό Γραμματέα και το, την ομάδα ελέγχου. Σύμφωνα με τον κανονισμό θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση έκθεση στα θεσμικά όργανα με τον αριθμό και το είδος των ελέγχων, της συστάσεις και τις δράσεις μετά από τις συστάσεις. Οπότε το θέμα της έκθεσης είναι οι δραστηριότητες των εσωτερικών ελεγκτών το 2008. Επίσης θυμίζω ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι ανεξάρτητη δραστηριότητα σχεδιασμένη κυρίως για να διασφαλίσει θέματα ελέγχων ε, διακυβέρνησης ορθής ε, ώστε να βελτιώνονται οι δράσεις των οργανισμών. Ε, επίσης αντικειμενικά θα πρέπει να αξιολογούνται τα τεκμήρια από τους εσωτερικούς ελεγκτές θα πρέπει να εντοπίζονται ευκαιρίες, ελλείψεις και υπάρχουν μετά δια, ε, συστάσεις με συνεχή διάλογο και επικοδομητικές διαβουλεύσεις που θα καταλήγουν σε συμφωνίες με τη διοίκηση σχετικά με τις προτάσεις και την υλοποίηση. Δέκα επαγγελματίες, δύο ε, βοηθοί προβλέπονται που λειτουργούν με επαγγελματισμό και βάση ε, τις προδιαγραφές που υπάρχουν. Το πρόγραμμα εργασίας για το 2008 καταρτίστηκε ε, με βάση προτεραιότητες τομέων σε σχέση με το προφίλ κινδύνου. Το 2008 το σύστημα ελέγχου έκανε πολλούς ελέγχους σε συγκεκριμένους επιχειρησιακούς τομείς και στο τέλος έγκριναν 17 εκθέσεις. Ορισμένα είναι σε μορφή προσχεδίου. Θα περιγράψω αρχίζοντας με δύο ελέγχους που καλύπτουν ε, τα τμήματα το, ένας οριζόντιος έλεγχος εξέτασε πόσο αποτελεσματικά ε, αντιμετωπίζει το Κοινοβούλιο τις εισερχόμενες ε, τιμολόγια μέχρι την πληρωμή τους. Η σημασία αυτής της διαδικασίας ε, υπογραμμίστηκε με αλλαγή κανόνων σε αρχές του 2008. Κάποιες, σε κάποιες περιπτώσεις ε, οι πιστωτές ε, βάζουν τόκους υπερημέρια αν καθυστερήσουν οι πληρωμές και τώρα υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις που μπορούν να αποφευθούν και μπορεί σε κεντρικό επίπεδο να απλουστευτεί η διαδικασία ενώ υπάρχει ο βασικός έλεγχος. Η έκθεση προτείνει μέτρα για να ε, ορθολογικοποιηθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία αποκέντρωση της ε, ευθύνης σε σχέση με την καταγραφή των δεδομένων και ηλεκτρονική επαλήθευση ε, ως επαλήθευση έγκρισης της πληρωμής θα πρέπει το θεσμικό όργανο έλαβε μέτρα ούτως ώστε να ε, βελτιώσει τον έλεγχο και να ε, εκπαιδεύσει τους χρήστες ακόμα. Μπορούν να γίνουν πολλά και υπάρχουν ε, απαιτούμενες δράσεις γι' αυτό. Οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι χρειάζονται δράσεις σε βασικούς τομείς, αναθεώρηση του κυκλώματος πληρωμής και επαλήθευση των ε, διαταγών πληρωμών ε, η δεύτερη, ε, το δεύτερο οριζόντιο τμήμα ε, αφορά τον εσωτερικό έλεγχο σε μακροπρόθεσμα, συμ, μακροπρόθεσμες συμβάσεις. Για την απαλλαγή του 2004, το Κοινοβούλιο είχε καλέσει από τη διοίκηση να βελτιώσει την παρακολούθηση των συμβατικών υποχρεώσεων μακράς διάρκειας ο έλεγχος, η καταλληλότητα των ελέγχων ε, δείχνουν όπου οι συμβάσεις ε, όποτε χρειαζόταν είχαν τις ε, κατάλληλες διατάξεις για τερματισμό και καταγγελία τους κλπ. Υπάρχουν και θέματα που πρέπει να, ακόμα να δούμε σε σχέση με τις συμβάσεις πλαίσιο μικράς διάρκειας που τώρα αποκλείονται, εξαιρούνται από τις προϋποθέσεις. Επίσης θα πρέπει οι όροι προϋποθέσεις να παρακολουθούνται ιδιαίτερα επειδή αλλάζουν οι τιμές και οι τεχνολογίες. Επίσης διαπιστώθηκε ότι θα υπάρχει δυνατότητα ορθολογικοποίησης ακόμη περισσότερο σε σχέση με την έκθεση σε κίνδυνο ε, και, να υπάρχουν και αυτόματες ρήτρες ανανέωσης. Παρακολουθούμε φέτος ε, τον έλεγχο αυτό. Περνώ σε άλλους τομείς που ελέγχθηκαν το 2008. Ε, εσωτερικός έλεγχος έχει μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική να ελέγξει όλους τους τομείς προσωπικών δαπανών μεμονωμένα δικαιώματα των υπαλλήλων ε, είναι το 20% ολόκληρων των, όλων των δαπανών και τις ε, πληρωμές ε, του, του μισθολογίου. Είδαμε το 2007, μετά δεύτερος έλεγχος το 2008 επικεντρώθηκε συγκεκριμένους τομείς κινδύνου που εντοπίστηκαν στον πρώτο έλεγχο. Θα έπρεπε να δούμε την κανονικότητα και νομιμότητα ε, των δαπανών και να δούμε ότι καταγράφονται σωστά στο μισθολόγιο των υπαλλήλων. Ο έλεγχος επίσης εξέτασε αν το νέο σύστημα μηχανογράφησης για τα προσωπικά δεδομένα ε, που λέγεται Streamline, προβλέπει αποτελεσματική διαχείριση σε αυτό το τομέα. Ο έλεγχος ε, επιβεβαίωσε την έκθεση στον κίνδυνο που είχε εντοπιστεί πριν και είδε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν, είχαν πραγματοποιηθεί κίνδυνοι. Υπάρχει <clears throat> μεγάλη δυνατότητα Βελτίωση εδώ, ε, γιατί υπήρχαν διπλές πληρωμές, ε, εδώ χρειάζεται συστηματική βελτίωση, ε, πιο δομημένες ανταλλαγές πληροφοριών, συχνότερες με άλλα θεσμικά όργανα, μειώνουν αυτούς τους κινδύνους, χρειάζονται πιο έγκαιρη παρακολούθηση των αλλαγών, επιδόματα τέκνων, νοικοκυριών κλπ. Χρειάζονται κριτήρια σε ό,τι αφορά την ημερήσια αποζημίωση, Επίσης ο έλεγχος είδε ότι η αντισταθμιστική αποζημίωση, το επίδομα αυτό το οποίο αντικαθιστούσε ένα παλιότερο δεν συνάδει με τους κανονισμούς για των υπαλλήλου. Υπάρχουν επίσης στο μοντέλο εξυγχρονισμού αδυναμίες που πρέπει να μας απασχολήσουν ε, κατεπηγόντως. Καλύτερη τεκμηρίωση, καλύτερος ε, επιμερισμός ε, καθηκόντων, ε, ακρίβεια δεδομένων. Για να δούμε όλα αυτά, ε, ο εσωτερικός έλεγχος συμφώνησε σε ένα πρόγραμμα δράσης με το προσωπικό που θα έπρεπε να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2009. Θα δοθεί συνέχεια και φέτος αυτό. Τώρα, άλλο βασικό θέμα ο εσωτερικός έλεγχος ε, δίνει προτεραιότητα στην παρακολούθηση και παροχή συμβουλών σε σχέση με το αποκεντρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου που είχε προβλεφθεί το 2003 από το Δημοσιονομικό Κανονισμό. Το πλαίσιο του 2003-2004 κάλυπτε όλα τα ε, τμήματα και τις υπηρεσίες του θεσμικού οργάνου. Ε, υπήρχαν συμπεφωνημένες δράσεις με δύο άκρα. Το ένα είναι να βελτιωθεί όλο το επίπεδο συμμόρφωσης με τα ε, επίπεδα στάνταρ ελέγχου και το άλλο είναι να ε, βελτιωθούν οι στόχοι σε σημαντικά σημεία ελέγχου. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου έκανε πολλές ελέγχους μετά για να δει σε ποιο βαθμό τα τμήματα και οι εσωτερικές υπηρεσίες εφάρμοσαν τις δράσεις. Ε, ποσοστό υλοποίηση ήταν περίπου 50% από ό,τι απεδείχθη. Η διοίκηση συμφώνησε αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα για τι εκκρεμεί δράσει 18. Θεωρήθηκαν κέρυες ε, γιατί αφορούσαν τομείς ε, και υψηλού κινδύνου. Το 2007 το IAS έκανε δεύτερη σειρά ελέγχων συνέχεια που ολοκληρώθηκαν το 2008. Ο 80% των αρχικών δράσεων έχουν υλοποιηθεί από ό,τι έδειξε το έλεγχος και οι περισσότερα τμήματα βελτίωσαν τα συστήματα εσωτερικής διαχείρισης και ελέγχου σημαντικά. Ο αριθμός μη ολοκληρωμένων δράσεων μειώθηκε από 18 σε 4 και αφορούν μεμονωμένο τμήμα. Όλες που θα είναι που είναι τώρα το αντικείμενο συγκεκριμένου ελέγχου ειδικού γι' αυτό. Τώρα πολύ σύντομα πάμε σε αριθμό άλλων τομέων που άρχισαν να μας απασχολούν το 2008 και τέλειωσαν το 2009 συνεχιζόμενη έλεγχη στις, ε, ε, στις δημόσιες προμήθειες βασικά στοιχεία της πολιτικής κτηρίων του Κοινοβουλίου σχεδιασμός, αξιολόγηση, διαχείριση των ε, ανάγκων που υφίστανται ε, και εφαρμογές ε, στον τομέα της μηχανογράφησης, τεχνολογίες της πληροφορίας. Εν συμπεράσματι, Το έργο του εσωτερικού ελέγχου το 2008 δείχνει σε σχέση με το συνολικό πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου τα περισσότερα τμήματα βελτίωσαν το επίπεδο της συμμόρφωσης με τους ελάχιστους στόχους ελέγχου των θεσμικών οργάνων, τα στάνταρ ελέγχου ε, και υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς ε, ε, κινδύνων στα τμήματα όπου ο έλεγχος έδωσε προτεραιότητα. Επίσης ε, υπάρχει αποδεδειγμένη πρόοδο σε κεντρικό επίπεδο σχέσεις με το, τους εξωτερικούς συνεργάτες, βελτίωση στην, στον καθορισμό προϋποθέσεων και αναγκών. Ε, είναι πολύ σημαντικό να δούμε ευαίσθητους τομείς, παραμένει αυτό προτεραιότητα, όπως και η ανάπτυξη και η υλοποίηση εναρμονισμένης προσέγγισης για τον εντοπισμό, καταγραφή, αξιολόγηση κινδύνων. Με χαρά σημειώνω ότι το 2010 η υλοποίηση αυτού του πλαισίου αποτελεί θεσμική προτεραιότητα. Το άλλο θέμα που θέλω να πω πριν κλείσω είναι ότι το έργο ελέγχου του 2008 κατέδειξε κατεπίγουσα ανάγκη καθορισμού προτεραιοτήτων εις ό,τι αφορά την ανανέωση ε, των ε, εντολών ε, που χρησιμοποιούν οι διατάκτες. Δεν έχω λάβει οδηγίες θα πρέπει να που ε, επηρέασαν την αντικειμενικότητά μου. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή, τους τον προκάτοχό του και τα τμήματα ε, των ε, διατακτών για την συνεργασία. Ευχαριστώ. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον ε, Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε αυτή τη θέση είμαι από τις 16 Μαρτίου 2009 ως εκ τούτου είναι η πρώτη μου παρουσία σε αυτή τη συνέλευση. Από το 2007 μέχρι 2009 ήμουνα διευθυντής του γραφείου του Προέδρου και προηγουμένως γενικός διευθυντής στην Επιτροπή Εσωτερικής Πολιτικής. Δεν έχω ασχοληθεί δηλαδή με το 2008 αλλά εφόσον αντικατέστησα τον προκάτοχό μου είναι καθήκον μου να το παρουσιάσω ορισμένες παρατηρήσεις. Καταρχήν σχετικά με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2008 και επίσης ε, να αναφερθώ στα θέματα που έφυξε ο κύριος Σαρμάς διότι ορισμένες απαντήσεις πρέπει να τις δώσω δημοσίως. Αναφέρθηκε σε τέσσερα θέματα. Θέλω να τον ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία μας, τη δυνατότητα επικομδοσίας δομητικών ανταλλαγών για το θέμα του οικειοθελούς συνταξιοδοτικού ταμείου, την ανταλλαγή σπουδαστών, τον συντελεστή πολλαπλασιασμού και ένα τέταρτο θέμα. Καταρχήν όσον αφορά την κατάσταση των βοηθών. Όπως ξέρετε, έχουμε ένα τελείως νέο σύστημα του υπολογισμού των βοηθών τόσο των ε, ε, ε, διεπιστευμένων όσο και των βοηθητικών και η βάση είναι η έκθεση απαλλαγής του 2006 που είχε καταρτιστεί και απετέλεσε την βάση για οκτώ ενιαία κριτήρια τα οποία πρότεινε ο Πρόεδρος και το Προεδρείο για την ε, κατάρτιση ενός νέου συστήματος και ε, τα, ε, οι αρχές αυτές υιοθετήθηκαν. Αν υπάρχουν λοιπόν πρόοδοι και ένα νέο σύστημα οφείλεται εις την εργασία της Επιτροπής σας στο παρελθόν και οφείλεται επίσης την προθυμία του Προεδρείου να χρησιμοποιήσει αυτές τις εργασίες σαν βάση για τις αποφάσεις τις οποίες έλαβε.

Ε, από ε, του έτους που ακολούθησε την εφαρμογή χρειάστηκε να επιλύσουμε διάφορα προβληματάκια στο σύστημα χωρίς να αμφισβητήσουμε το συνολικό σύστημα. Αναφερθήκαμε στα έξοδα ταξιδίου ή στις προκαταβολές των βοηθών ε, ή παραδείγματος χάρη βοηθούς οι οποίοι μετά από δύο μήνες ασθενείας ε, πρέπει να έχουν μία σωστή περίθαλψη, το ίδιο και ε, για τους βουλευτές και τα μέλη των οικογενειών τους οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ε, επίδομα ενός μηνός το οποίο μεταφέρεται για τα έξοδα βοηθού από το ένα έτος στο άλλο για να αποφύγει κανείς ε, δαπανηρούς ε, τοπικούς βοηθούς κατά τρόπον ώστε να καλύπτονται κατά αποκοπήν τα έξοδα ταξιδίου του αρμοδίου. Όσον αφορά το, συνταγματικό, το, το συνταξιοδοτικό ταμείο. Ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις διότι το 2009 στην αρχή του χρόνου διαπιστώσαμε ότι είχε ένα μεγάλο κενό το ταμείο, λογιστικό ε, κενό, το οποίο βέβαια δεν γνωρίζουμε πόσο είναι στην πραγματικότητα, γιατί θα το γνωρίζουμε μόνο αν το ταμείο, οπότε το Προεδρείο αποφάσισε να Θέση με το παρελθόν να μην ζητήσει επιπρόσθετες ε, συνδρομές από τους ε, τρέχοντες ευρωβουλευτές ε, αλλά να κάνει αλλαγές στην μέχρι του ρύθμιση του Ταμείου και ε, να μεταφέρει το έτος ε, εξόδου από τις ε, συνδρομές από τα 60 στα 63 χρόνια και ήταν ένα πρώτο μέτρο που λήφθηκε για να αποφευθεί η διαρροή κεφαλαίων και να εξασφαλιστεί η ρευστότητα. Υπήρξαν και άλλα μέτρα τα οποία ελήφθησαν δεν ανελήφθησαν νομισματικοί κίνδυνοι και η νομική υπηρεσία διευκρίνησε ότι διαμέσου των ετών και με την στενή διασύνδεση Κοινοβουλίου και Συνταξιοδοτικού Ταμείου εάν κάποια στιγμή τελείωναν οι πόροι του Συνταξιοδοτικού Ταμείου το Κοινοβούλιο δεσμεύεται να καλύψει τις υπόλοιπες συντάξεις των Ευρωβουλευτών πράγμα το οποίο είναι μία διευκρίνηση μία απόφαση που έλαβε το Προεδρείο και αντικατοπτρίζει δημοσιονομικά και την πραγματικότητα διότι αν υπάρχει μία τέτοια κατάσταση θα πρέπει να το γνωρίζει κανείς στο τέλος του έτους να είναι μία διάφανη διαδικασία για να γνωρίζουμε τι ποσά ενδέχεται να χρειαστεί να καλυφθούν στο μέλλον. Όσον αφορά την αποζημίωση ταξιδίου υπήρξε ε, καλή και επικοδομητική συζήτηση με το ελεγκτικό συνέδριο το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η μέχρι τούδε ρύθμιση για τους υπαλλήλους δεν ε, έχει λάβει επαρκώς υπόψη την ε, ιδιομορφία του Κοινοβουλίου διότι ένα μέρος των ε, εργαζομένων έχουν έδρα στις Βρυξέλλες, ένα μέρος στο Λουξεμβούργο και το ίμιση ε, αυτών που ε, διαμένουν στο Λουξεμβούργο πρέπει μία φορά το μήνα να φεύγουν από τα σπίτια τους να πάνε στο Στρασβούργο το ίδιο ισχύει και ε, για τους διαμένοντες στις Βρυξέλλες και εξαρτάται βέβαια από την ερμηνεία του κανονισμού είχαμε θεωρήσει ότι αυτό δεν είχε γίνει επαρκώς αντιληπτό εις ε, από το ελεκτικό συνέδριο και στον επόμενο κανονισμό προσωπικού θα πρέπει να διευκρινιστεί για να ξεχωρίζει κανείς τα απλά ταξίδια ε, και ε, από τα συνήθη μεταξύ Βρυξελών, Στρασβούργου και Λουξεμβούργου και αυτό μπορεί ίσως να επιτευχθεί μέσω ε, της Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Υπηρεσίας. Ήδη έχουμε προσαρμόσει ε, το σύστημά μας για να λάβουμε υπόψη μας αυτή τη ρύθμιση και έχουμε λάβει υπόψη και ορισμένες κρίσεις που είχαν αναφερθεί παραδείγματος χάρη όσον αφορά την αποπληρωμή κατά αποκοπή μια ημέρας εάν ξεκινάει κανείς πολύ νωρίς ή γυρίζει σπίτι του αργά τη νύχτα. Ε, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής μία ενιαία αντιμετώπιση από τα διάφορα θεσμικά όργανα και ε, σε αυτή την περίπτωση χρειάστηκε να προσανατολιστούμε προς ε, την μέθοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία εντωμεταξύ είχε αλλάξει το σύστημά της. Δηλαδή στην αρχή της διαδικασίας ε, την τωρινή μέθοδο δεν τη θεωρούσε σωστή και χρησιμοποιούσε διαφορετικό σύστημα. Άρα τώρα πρέπει να υπάρχει μία διευκρίνηση για την ενιαία αντιμετώπιση και όταν θα υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση θα καλύψουμε ε, τα θέματα αυτά. Αυτά όσον αφορά την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Θα ήθελα όμως να πω ακόμη μερικά λεπτά ε, ε, σχετικά με τις εμπειρίες μου στο Κοινοβούλιο από όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου στις 16 Μαρτίου διότι ε, όταν ε, ε, προετοιμάζεται κανείς για μια τέτοια θέση πρέπει να ασχοληθεί ενεργητικά με το οργανόγραμμα και με τις διεργασίες. Γι' αυτό και εγκαίρως διαπίστωσα ότι πρέπει να ενεργήσουμε επιγόντως στον τομέα της ασφάλειας, των κτηρίων και του προσωπικού. Εγώ ε, ξεκίνησα τα καθήκοντά μου 16 Μαρτίου, 23 Μαρτίου. Έκανα μία πρόταση στο Προεδρείο για αναδιάρθρωση σε τομείς, την οποία υιοθέτησε το Προεδρείο στην 1η Απριλίου. Καταρχήν γιατί στον τομέα ασφαλείας το Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί πέραν των 800 εξωτερικών συνεργατών. Γνωρίζουμε όλοι ότι όταν υπάρχουν προβλήματα τα οποία έχουν σχέση και με κίνδυνο και με απώλεια της, του κύρου του Κοινοβουλίου και γι' αυτό το Προεδρείο αποφάσισε να καταρτήσει μία διεύθυνση ψάχνουμε αυτή τη στιγμή έχουμε προκηρύξει για έναν διευθυντή όχι μόνο εσωτερικό συνεργάτη αλλά ίσως και έξω θα υπάρχει ένας γενικός διευθυντής λοιπόν και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε και την εσωτερική μας εμπειρία μέσω άλλων διοικητικών υπαλλήλων. Πέραν αυτού σε πολλά θέματα οι δομές μας δεν ανταποκρινόντουσαν στις ανάγκες, δεν είχαμε δώσει αρκετή σημασία εις ε, την ε, ε, συντήρηση διότι ενδέχεται σε ένα το οποίο είναι νέο αλλά φαίνεται να γερνάει και είχαμε ένα κραυγαλαίο παράδειγμα με την οροφή της Ολομελίας στο Στρασβούργο και αντιλαμβάνεται τι μπορεί να συμβεί αν δεν δώσουμε τη δόση προσοχή σε αυτό το θέμα. Αυτό τώρα έχει διασφαλιστεί εις την οργάνωση, δηλαδή άλλες είναι οι νέες ενέργειες και άλλες είναι οι ενέργειες συντήρησης. Ε, υπάρχει και κεντρικό, μια κεντρική οικονομική διαχείριση για τα ποσά τα οποία διαπιστώσαμε ότι κακώς δαπανούνται και ε, η Ολομέλεια δέχτηκε το πρόγραμμά μας για μία τριετία να χρησιμοποιήσουμε επιπλέον εμπειρογνώμονες κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την ε, εξωτερική εμπειρία και αυτό που είναι επίσης σημαντικό είναι να λάβουμε υπόψη ότι έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα στο Λουξεμβούργο που προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε όλα τα κτίρια σε λιγότερες μονάδες. Ε, ε, όσον αφορά το θέμα του δημοσιονομικού ελέγχου είναι βασικό να πούμε ότι υπάρχει μία διεύθυνση η οποία αναφέρεται στα ατομικά δικαιώματα και στην εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού κατά τρόπον ώστε να υπάρχει ενιαία εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού διότι είπε ο ελεγκτής ότι 20% του, των αμοιβών του προσωπικού προέρχεται από προσόντα τα οποία θα πρέπει να έχουν εξακριβωθεί. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μία εφαρμογή και η Γενική Διεύθυνση η οποία έχει τα μεγαλύτερα έξοδα δεν είναι η Γενική Διεύθυνση των κτηρίων αλλά προσωπικού. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να σας αναφέρω και που αντικατοπτρίζεται και στην έκθεση είναι ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να υπάρχει μία ισορροπία μεταξύ του τι γίνεται εσωτερικά με τις εσωτερικές μας δυνάμεις και τι ε, πρέπει να ανατεθεί ε, ως υπεργολαβία. Είναι θέμα ισορροπίας στο κάθε δεδομένο τομέα διότι πιστεύω ότι στον τομέα της ασφαλείας των κτηρίων και στην τεχνολογία πληροφορικής ε, κάνουμε υπερβολική ανάθεση εξωτερική και από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν άλλοι τομείς όσον αφορά τις γλώσσες, τη μετάφραση όπου ίσως υπάρχουν επιπρόσθετες δυνατότητες ιδίως αν δούμε τους αριθμούς για το κόστος της ε, μετάφρασης το οποίον διαπιστώνουμε βλέπουμε ότι η εσωτερική μετάφραση κοστίζει τρεις φορές περισσότερο από την εξωτερική. Βεβαίως θα είναι και διαφορετική σε η εσωτερική εξωτερική μετάφραση από αυτή την οποία θα μας προσφέρουν οι εξωτερικοί συνεργάτες. Ε, είναι ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε με τους ε, ελεγκτές, επίσης το, την πληροφορική, το σωστό σύστημα που πρέπει να εφαρμοστεί και εγώ εξεπλάγει ότι δεν υπάρχει ένα τμήμα το ε, οργανόγραμμα που να ασχολείται με την οργάνωση του προσωπικού. Ε, ξέρω ότι ο εισηγητής ενδιαφέρεται για ορισμένα θέματα όπως είναι οι εξωτερικές αγορές. Μας είπε ο ελεγκτής ότι οι ε, δημόσιες αγορές είναι πολύ σημαντικές. Ένα θέμα έχει ολοκληρωθεί, αλλά αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται. Αλλά νομίζω ότι ήδη μπορούμε να καταλήξουμε σε ορισμένα συμπεράσματα. Διαπιστώσαμε αδυναμίες οι οποίες ε, οφείλονται σε όλη την αλυσίδα από τον ε, προγραμματισμό στη συγκεκριμένη διατύπωση, στην αξιολόγηση και στην ε, επικοινωνία. Το σημείο εκκινήσεως του, προβλήματος είναι στον προγραμματισμό. Έχουμε δυναμίες προγραμματισμού των δραστηριοτήτων μας και δεν είμαστε ε, επαρκώς ακριβείς εις ε, τις προκηρύξεις μας. Αυτά είναι θέματα που δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο τομέα αλλά καλύπτουν όλη την οργάνωση. Από το καλοκαίρι έχω ξεκινήσει ε, ένα διοικητικό πρόγραμμα εργασίας 2010-2011 όπου θα συμμετάσχουν επί δυόμιση χρόνια όλες οι γενικές διευθύνσεις και ελπίζω ότι κατά αυτό αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να επιλύσουμε αυτές τις αδυναμίες. Πρέπει όμως να υπάρχουν αντίστοιχε προγραμματισμοί και στο πολιτικό τομέα, στην πολιτική των κτηρίων και στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας και το Προεδρείο δεσμεύτηκε προς την Επιστροπή Προϋπολογισμού μέχρι το Μάρτιο να διατυπώσει μία μεσοπρόθεσμη στρατηγική για τα κτίρια και ε, για το θέμα της οργανώσεως γενικότερα. Μπορώ να επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες για τα κτίρια, αλλά ίσως δεν είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή. Επίσης, όσον αφορά τη διαχείριση του κινδύνου, ε, ήταν αμφιλεγόμενο εάν χρειαζόταν ένα risk management αλλά μάλλον που έπρεπε να εδρεύει είτε στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών είτε της Προεδρίας την Οικονομική Γενική Διεύθυνση θα ε, μπορούσε κανείς να δώσει την εντύπωση ότι αναφερόταν ε, σε ε, οικονομικούς κινδύνους ενώ δεν θέλουμε μόνο να αποτρέψουμε οικονομικούς κινδύνους κινδύνους αλλά και μη οικονομικούς κινδύνους. Αν γινόταν ε, αντιθέτως εις ε, το Προεδρείο, ε, στην Προεδρία θα τόνιζε κανείς περισσότερο την ασφάλεια των ατόμων και τον κίνδυνο των κτηρίων. Επειδή υπήρχαν αυτές αυτά τα ερωτηματικά αποφάσισα να αναλάβω εγώ προσωπικά την ε, το τμήμα αυτό και να αναλάβω την ευθύνη ε, στο επίκεντρο διότι σημασία έχει να επιλύσουμε τους οριζοντίους κινδύνους ε, εάν δηλαδή ε, υπάρχει ένας μάνατζερ κινδύνου ο οποίος αξιολογεί τον κίνδυνο και θα αναφέρεται κατά τρόπον ώστε να μπορεί να ε, μειώσει τους κινδύνους να τους αποτρέψει και να βρει λύσεις. Είναι μία προτεραιότητα για το 2010 να καταρτήσουμε αυτό το σύστημα το οποίο θα λειτουργήσει σωστά μόνο αν υπάρχει ένα δίκτυο δηλαδή αν εμπλακούν όλες οι γενικές διευθύνσεις κατά τρόπον ώστε να έχουμε μία γενική ε, ε, συγκέντρωση των πληροφοριών όλες οι γενικές διευθύνσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στο έργο αυτό και σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε τον Γενικό Γραμματέα και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Στάις, τον εισηγητή. Ehm, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την εισαγωγή. Βέβαια υπάρχει κάποιο, ε, πρόβλημα χρόνου, αλλά επειδή ε, ε, θα, γι' αυτό θα περιοριστώ στα σημαντικά. Πολλές ερωτήσεις που θα ήθελα να θέσω δεν θα προλάβω. Θα επικεντρωθώ στα σημαντικότερα. Ε, η απαλλαγή είναι σημαντικό πράγμα. Δηλαδή απαλλάσσουμε τις ευθύνης ε, κάποιους. Πρέπει να το κάνουμε αυτό με βάση στέρεη. Γι' αυτό ανησυχώ. Παρά τα λόγια από το ελεγκτικό συνέδριο, από τον κύριο Γκάλβιν, παρά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα και των προκατόχων τους. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, τώρα δουλεύουμε με το νέο δημοσιονομικό κανονισμό και υπήρξαν διοικητικές μεταρρυθμίσεις Τώρα δε έχουμε ένα σύστημα αποκεντρωμένης δημοσιονομικής διαχείρισης. Η έννοια του εσωτερικού ελέγχου εδώ παίζει ρόλο κλειδί. Δεν είναι το μοναδικό στοιχείο, αλλά είναι θεμελιώδες. Το κοίταξα αυτό στο δημοσιονομικό κανονισμό για να δω, να δω τι λέει. Στο άρθρο 16.7 ε, αναφέρει τι περιμένουμε από ένα σύστημα IAS, δηλαδή σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σε σχέση με τους διατάκτες που μετά θα πρέπει να τα δουν όλα αυτά. Στο άρθρο 67 λέει ότι ε, στη ετήσια έκθεση θα τα Τέλο πάντων, αναφέρεται ότι πρέπει να βελτιώσουν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και αυτό ήταν ένα σημαντικό ερώτημα για μένα. Εξεπλάγει, κύριε Γενική Γραμματέα, όταν διάβασα την απάντηση στην ερώτησή μας 4, 2 στις 6 και 7 σελίδες γιατί εκεί ομολογείται ότι δεν είναι όλοι οι διατάκτες ε, διατεθειμένοι και δεν καλούνται να υποβάλουν έκθεση σε σχέση με τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου. Λέτε ότι είναι κάποιοι που πράγματι υποβάλλουν έκθεση. Όχι όλοι όμως και αυτό είναι ανησυχητικό. Πώς είναι αυτοί, κανένας δύο, τρεις, τέσσερις ε, ε, υποβάλλουν έκθεση όπως πρέπει και οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα. Οι μισοί κάνουν, οι άλλοι δεν κάνουν. Πρέπει να τα ξέρουμε αυτά λεπτομερέστερα για να ξέρουμε αν όντω υπάρχει αυτή η στερεή βάση που σας έλεγα και να δούμε αν οι αιτήσιες εκθέσεις των διατακτών είναι σωστές. Βέβαια δεν είστε υπεύθυνο για το 2008, το ξέρω, αλλά οι απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσεις μας ε, δεν είναι πλήρης. Δηλαδή ήδη τώρα ε, προσπαθήσατε να λάβετε τα ανάλογα μέτρα, οι διατάκτες είναι υποχρεωμένοι να φροντίσουν για το μέλλον τόσο ώστε ε, να εφαρμόζεται πραγματικά το 2009 το άρθρο 67 και προς το ελεγκτικό συνέδριο. Λέτε ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι καλό. Βλέποντας όμως ότι μια σειρά διατακτών δεν το εγκολπώνονται και δεν το εφαρμόζουν, ε, τότε πώς θα έχουμε στερεή βάση. Δεύτερο στοιχείο. Η δήλωση αξιοπιστίας που πρέπει να δώσετε ως Γενικό Γραμματέας. Ο προηγούμενος, ο κ. Ρόιμερ, το έκανε το Μάρτιο για το 2008 και λέει κάποια στιγμή στην επιστολή του και το αναφέρω στα αγγλικά ε, καταρτίζει την ετήσια έκθεση με βάση τα στοιχεία από το διατάκτη. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Δεν γίνεται εκεί καμία παρατήρηση στο, στην επιστολή του κυρίου Ρόμερ. Δεν λέει ότι ακολούθησαν όλοι οι διατάκτες ε, τις προδιαγραφές που θέτει ο δημοσιονομικός κανονισμός. Δεν ήλεγξαν την ε, ε, αποτελεσματικότητα. Είναι μια δυναμία στο σύστημα που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Ο πρώην γενικός γραμματέας συνεχίζει την επιστολή του και παραθέτω λαμβάνει υπόψη ότι κανένας διατάκτης της δηλώσεις του δεν έχει προβεί σε περιορισμούς. Μπορεί να μην έχει, κάνει, να μην έχει βάλει κάποιους περιορισμούς, ε, ε, κάποιους διατάκτης, αλλά το γεγονός ότι δεν έγινε αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε και λόγος να μην το κάνει. Και αυτό είναι μια δεύτερη αδυναμία του συστήματος. Και στην ε, έκθεση απαλλαγής, εγώ θα το τονίσω αυτό, θέλω δεν να ξέρω ποια είναι η γνώμη σας και η γνώμη των συναδέλφων σας Δηλαδή, έχουμε μια ετήσια έκθεση και μια δήλωση και αυτό είναι σαν έκθεση διαχειριστική, δηλαδή αναφέρεται τι έγινε, ε, αναφέρεται στο ε, σύστημα εσωτερικού ελέγχου αλλά από την άλλη δεν υπάρχει ένα αντίβαρο ή ένα πρώτο-δεύτερο δείγμα ελέγχου. Στην ερώτηση 4-7 το λέω αυτό. Δεν πρέπει να σκεφτούμε μήπως ε, θα πρέπει να έχουμε μια προνοιακή λειτουργία, να υπάρχει δηλαδή κάποιος που θα παρακολουθεί την όλη διαδικασία και θα βλέπει θα, ε, αν υπάρχει, θα, θα λειτουργεί και ως αντίβαρο και θα φροντίζει για την καλή λειτουργία του συστήματος. Θα μπορούσα να πω περισσότερα πράγματα, αλλά περιορίζομαι σε αυτά που είναι σημαντικά και για σας, ε, κυρία Γενική Γραμματέα. Ε, σύντομα θα κληθείτε να δώσετε την πρώτη δήλωση αξιοπιστίας. Και βεβαίως ε, εδώ μιλάμε για πολλά χρήματα, 1,5 δις ευρώ. Και νομίζω ότι μαζί θα πρέπει να προβληματιστούμε σχετικά με την ενίσχυση, δυνατότητα ενίσχυσης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, τόσο ώστε να υπάρχει ένα αντίβαρο. Όταν εσείς δηλαδή υπογράφετε τη δήλωση αξιοπιστίας σας, να μην το κάνετε τυπικά, αλλά επειδή όντω υπάρχει μια στέρεη βάση για να γίνει. Έτσι μπορούμε να αρχίσουμε, πέρα από πολλά άλλα που πρέπει να γίνουν. Είναι τρίτη φορά που είμαι εισηγητής για την απαλλαγή του Κοινοβουλίου έχετε διαβάσει και άλλες εκθέσεις, ξέρετε τις απόψεις μου, ξέρετε ότι με μεγάλη σοβαρότητα ασχολούμαι και με, και με ε, περιδικαίου αίσθημα ασχολούμαι με όλα αυτά. Ε, όμως είναι πολύ σημαντικό το θέμα των εσωτερικών ελέγχων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, θα δώσω το λόγο στο Γενικό Γραμματέα, αλλά σας υπενθυμίζω σε όλους ότι θα, τελειώσουμε στις 7. 7 και 4 μου έχουν δώσει μέγιστο όριο, γιατί ζήτησα λίγο παραπάνω χρόνο. Μέχρι 7 και 4 λοιπόν. Δεν θα ξεπεράσουμε τι 7 και 4. Äh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις του εισηγητή που ήταν σωστές. Καταρχήν, βεβαίως, θα πρέπει να συμφωνήσουμε, να διαπιστώσουμε ότι ο κάθε ένας ο οποίος κάνει αυτή τη δήλωση ε, αναλαμβάνει ε, την πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση του τομέα του και αυτή ήταν η ουσιαστική αλλαγή την οποία κάναμε μετά από το 1998 όλα αυτά νομίζω ότι σωστά τίθεται η ερώτηση, δηλαδή αν δεν μπορούμε να βελτιώσουμε το σύστημα. Και θα ήθελα να συμφωνήσω ότι η έκθεση πρέπει να είναι πιο απλή και αυτό που είναι πιο σημαντικό πρέπει να είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων και ο Γενικός Γραμματέας πρέπει να έχει πιο, πιο στενό διάλογο με τους υπευθύνους προτού καταρτήσουν αυτή τη δήλωση διότι οι οδηγίες για τους εντεταλμένους διατάκτες ε, για το 2009 ήταν πολύ πιο αυστηρές από το 2008 άρα ελπίζω ότι τα προβλήματα τα οποία θίξατε δεν πρόκειται να υπάρξουν ε, τόσο το 2009. Βεβαίως, ο, ο, ο, ο βασικός διατάκτης δεν έχει μόνο αυτή τη δυνατότητα μπορεί να προβεί σε συζητήσεις μπορεί να χρησιμοποιήσει ε, την, ε, ε, την πληροφορική μπορεί να χρησιμοποιήσει τα μέσα του εσωτερικού ελέγχου και ελεγκτή. Αλλά συμφωνώ, το θέμα αυτό πρέπει να είναι ε, ε, να δίνει μία πιο σαφή ε, εικόνα, να είναι συγκρίσιμα, πιο λεπτομερή, και να μπορούν να με βοηθήσουν για να καταρτήσω στο τέλος τη δική μου δήλωση. Ευχαριστώ. Άλλη, άλλο ερώτημα κύριε Στάς. Δίνω το λόγο τότε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Ευχαριστούμε για τις πολλές απαντήσεις που ελάβαμε. Διευκρινίζω. Όταν ε, υπάρχει ένα κτίριο πληρώνουμε το 30% περισσότερο από ό,τι θα ήταν η κανονική τιμή αγοράς. Στην περίπτωση του Κοινοβουλίου συμβαίνει αυτό. Είναι αλήθεια αυτό και πώς πρέπει να διερευνηθεί. Επίσης, για την ε, πολιτική των κτηρίων. Στο Στρασβουργό είχαμε πρόβλημα μιάντου και έγιναν οι επισκευές. Όμως αγοράστηκε από το Δήμο του Στρασβούργου το κτίριο αυτό. Δύο εκατομμύρια πλήρωσε ο Δήμος του Στρασβούργου παρόλο που το συνολικό κόστος ήταν τρία εκατομμύρια κανονικά θα έπρεπε να τα πληρώσουν όλα. Γιατί πλήρωσαν μόνο ένα μέρος. Επίση όταν έπεσε η σκεπή, η οροφή, ο Δήμος του Στρασβούργου που πούλησε το κτίριο δεν ε, ε, σύρθη στο δικαστήριο όπως ε, θα έπρεπε κανονικά. Νομίζω ότι ε, και ο πολιτής ε, πλήρωσε. Επίσης, ε, σε άλλα κτηρία αργούν πολύ, καθυστερούν οι κατασκευές, ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Εν τω μεταξύ το πολιτικό κλίμα λένε ότι έχει αλλάξει. Όμως το, στο κέντρο πληροφοριών δεν είναι δικαιολογία γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Και πώς θα συνδεθούν τα δύο. Επίσης, ε, την καλύτερη μέρα ας πούμε ε, παρακολουθούν τη τηλεόραση του Κοινοβουλίου 10.000 ε, συνήθως 5.000 αν αφαιρέσουμε τους βοηθούς και τα μέλη του Κοινοβουλίου είναι δηλαδή μερικές χιλιάδες ε, θεατές και έχουμε 500, 500 εκατομμύρια στην Ευρώπη δεν ε, αποδίδει επένδυση δηλαδή. Επίσης, ε, για το, τις θερινές διακοπές για σκι, λέει στο, στην εφημερίδα ο, κάποια στιγμή ότι εμείς ε, παίρναμε επιδόματα ή πληρωμές για να κάνουμε χειμερινές διακοπές για σκι. Αλήθεια είναι αυτό γιατί δεν πρέπει, κάτι πρέπει να κάνουμε τόσο ώστε αυτές να μην είναι συζητήσεις οι οποίες ζημιώνουν το, το κύρος του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Στο θέμα των κτηρίων. Για τα κτίρια, όσον αφορά τις Βρυξέλλες, βεβαίως, αντικειμενικά, είμαστε πάντοτε σε δυσχερή θέση διότι δεν θέλουμε να έχουμε ένα κτίριο που είναι στην άλλη άκρη της πόλεως ή που δεν είναι εύκολης πρόσβασης και επίσης για λόγους κόστους. Για την γενική οργάνωση χρειαζόμαστε κτίρια τα οποία να μπορούν να είναι κοντά στο ισχύον σύστημά μας. Αν δεν είμαστε δεμένοι με αυτά τα κτίρια δεν θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε και τα Και αυτό μας φέρνει σε δύσκολη θέση όταν διαπραγματευόμαστε γιατί υπάρχουν λίγα κτίρια τα οποία για μας μπορούν να είναι ενδιαφέροντα για να τα αγοράσουμε. Άρα ε, μπορούμε αυτά να τα περιγράψουμε εύκολα. Όσον αφορά τον αμίαντο, όπως είπατε πολύ σωστά, ε, πήραμε 2 ε, εκατομμύρια ευρώ από, το Στρασβούργο, από την πόλη του Στρασβούργου, τα οποία βέβαια είναι λιγότερα από τα 3 εκατομμύρια. Όσον αφορά το κέντρο πληροφοριών, ε, είναι ένα μοναδικό κέντρο επισκεπτών στην Ευρώπη, καταρτίζεται σε ένα κτίριο το οποίο στην αρχή δεν είχε προβλεφθεί για κτίριο επισκεπτών και από ό,τι κατάλαβα επρόκειτο να γίνει γκαράζ. Πράγμα βέβαια το οποίο δεν διευκολύνει την κατάσταση και υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις διότι η προκήρυξη δεν λειτουργήσε καλά του διαγωνισμού και ξέρετε ποιοι είναι οι, κα... οι κανόνες. Εάν επαναληφθεί ο διαγωνισμός χάσαμε ήδη μισό χρόνο. Αλλά ε, Βέβαια ε, η προκήρυξη του διαγωνισμού πρέπει να προεξοφλεί ε, μια επιτυχή περαιτέρω προκήρυξη και άρα έχουμε να λύσουμε διάφορα προβλήματα και όσον αφορά τη χρήση των πολυμέσων νομίζω ότι κάτι χρειαζόμαστε και πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει ε, το, η συνθήκη της Λισαβόνα τώρα. Δηλαδή δεν μπορούμε ε, να σεβόμαστε τις αρχές που υπήρχαν ε, πιο προ-Λισαβόνας. Πρέπει να ενημερώσουμε τα στοιχεία και αυτό επίσης έχει οδηγήσει σε ορισμένες καθυστερήσεις. Όσον αφορά την τηλεόραση του Κοινοβουλίου, έχω εδώ αριθμούς ή στο φάκελο τους οποίους διευκρίνησα όσον αφορά τις διακοπές για σκι Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου ένα ποσό το οποίο διαθέτει το Κοινοβούλιο κάθε χρόνο και επιτρέπει στο Συμβούλιο του Προσωπικού να οργανώσει ένα όγκο μεταξύ 150 ε, ε, και 200 χιλιάδων ευρώ για δραστηριότητες πέραν των οργανώσεων οργανωτικών θεμάτων, για κοινοτικέ ε, ε, ε, δραστηριότητες και μόρων. Και το Συμβούλιο Προσωπικού αποφασίζει πώς θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά. Δεν μπορεί να παρέμβει ούτε η διοίκηση ούτε ο Γενικός Γραμματέας. Διαθέτουμε αυτά τα χρήματα. Πέρυσι διατέθηκα σαν για διάφορες δραστηριότητες μεταξύ των οποίων ήταν και ένα ταξίδι για σκι, άλλες ε, ε, εξωτερικές δραστηριότητες για τα παιδιά ε, κατά το, έκτος, το έτος 2008 που συζητάμε τώρα 72 παιδιά ενεπλάκησαν, πήγαν δηλαδή για σκι και